Colleagues. Συνάδελφοι. Can I bring the meeting? Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και να πιάσουμε το επόμενο σημείο στην μιλήσει διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Κατά πρώτον, να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των συντονιστών από τις 14 Οκτωβρίου κυρίως για τα σκάφη των εσωτερικών πλωτών οδών δύο εκθέσεις για εισηγητές Η γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού και δημοσιονομικού κανόνε που θα ισχύουν στον γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισηγητή από την έκθεση προπολογισμών. Και επίση, διορισμός διευθυντή για, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Και καμία απόφαση των συντονιστών για τα υπόλοιπα. Οι ετήσιοι λογαριασμοί για το ΣΕΖΑΡ και τον ε, Οργανισμό των Συμπυροδρόμων από κοινού από το ΕΛΚ για όλους τους οργανισμούς, για όλους τους, ε, συγγνώμη, τους οργανισμούς. Ως προς τις οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι μια αντιπροσωπεία 6 μελών θα πάνε στη Μαδέρα την εβδομάδα που ξεκινάει 14 Μαρτίου, 14 με 20, είναι η μόνη εβδομάδα που έχουμε την ευκαιρία. Δεν θα γίνουν ακροάσεις το πρώτο τρίμηνο του 2014. Επίσης, λάβαμε μια έκθεση επιτροπολογία και έπειτα για τι συνεδρίε των συντονιστών τη χθεσινή οι μία γνωμοδότηση για το σύστημα εναλλαγής, το ΕΛΚ ανέλαβε για το ETS Οι συντονιστέ θα αποφασίσουν στη συνέχεια, καμία απόφαση για τα υπόλοιπα και θα σας μοιραστούν και τα ενημερωτικά κείμενα. Για τι διαστικές ε, περιοχές, ε, μεταφορές σε από κέντρες περιοχές αποφασίσαμε παρουσίαση τη μελέτη σε μια από τι επόμενε συνεδριάσεις τη επιτροπή μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το προβλέψουμε σε μια ε, από τι επόμενε συνεδριάσεις. Άρθρο 51 για τον ΑΕΔΙΣ απόφαση των συντονιστών να απορριφθεί η αίτηση από την Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά συμφώνησαν να εφαρμοστεί το άρθρο 50 για τα πρώτα δύο εδάφια του άρθρου 8. Κοινέ αρμοδιότητες για τα εναπομείναντα. Επίσης, ζητήθηκε από τη Γραμματεία να διερευνήσει τη δυνατότητα να οργανωθεί ακρόαση Επίσης ανταλλαγή απόψεων για την αεροπλοεία. Απόφαση επιτροπολογίας. Αυτά από τη χθεσινή ε, συνάντηση των συντονιστών και την προηγούμενη. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά. Εάν όχι, <clears throat> να προχωρήσουμε απευθείας. Ψηφοφορίες. Έχετε όλες τις κάρτες σας για τα μηχανήματα. If you have your cards Εάν έχετε τις κάρτες σας, να περάσουμε σε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Αυτό για να δούμε ότι το ΕΛΚ δεν έχει περισσότερα μέλη. At Προς στιγμή είναι όλα καλά. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Ωραία λοιπόν, ως εδώ όλα πάνε καλά. Απλώς τεστ ήταν αυτό. Κι άλλο τεστ λοιπόν, για να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι υπεράριθμο το ΕΛΚ. Ξανά ψηφίζουμε. It'll be crazy if somebody else is over now, won't it, when you're Θα ήταν παράλογο να είναι οι υπόλοιποι υπεράριθμοι. Εντάξει, σωστά είμαστε. Ξεκινούμε. Πρώτα απ' όλα θα βάλω το τσάι μου στο φλιτζάνι. Ολοκληρωμένη αγορά παράδοση δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισηγητή ο κ. Νταντνά. Τροπολογία 1. Ξεχωριστή ψηφοφορία όπω τη ζήτησε το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα. Αναγνωρίζει τη σημασία και ποιότητα των υπηρεσιών διανομή. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα πρέπει να το ψηφίσουμε. Ωραία λοιπόν. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 Λίχτεμπεργκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τρίτη τροπολογία. να απαντήσω. Πέρας. 16 υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται συμβαστική σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 24 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία να ψήφισαν άπαντες πέρασε εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε για τον 25. Έψηφσαν άπαντες. πέρας. Εγκρίνεται. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. F. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να, ελάξουμε, να ψηφίσουμε on μπλοκ τη 48 με 55. Όχι, 50 διαφέρει. 48 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Έψηφισαν άπαντες. Πέρας. 37 υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται και μάλιστα ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Νταντά. Ελπίζω όταν κοιτάξουμε και το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο να φανεί αυτή η ομοφωνία και στη συνέχεια. Επόμενη. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, κυρία Μάισνερ. Κύριε Κουν, μισό λεπτό να βρω τα ακουστικά μου. Για ξεκινήστε. Υπάρχουν κάποιε τροπολογίες που τις επέβαλα εγώ ίδιο για τι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Η τροπολογία 209 και 212. Θα τις αποσύρω. Διότι η διατύπωση είναι ακόμη πιο συγκεκριμένη σε σχέση με αυτή που προτείνει η συγκεκριμένη κυρία Μάισνερ. 209 και 212. Thank you for that, right. Εντάξει, θα το σημειώνουμε. Ξεκινάμε. Η πρώτη είναι γλωσσική, οπότε πάμε στην 11 του εισηγήτριας. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ ...82 ως προσθήκη. Κούν. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Νομίζω απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. 82. 82 ως προσθήκη. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Ξανά. 83 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Envy. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Το κυρίου Κομιτσάκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι γκρίθηκε, αλλά να ελέγξουμε. 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Έψηφαν άπαντες. Πέρας. 27 υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. Ελάτε, σηκώντε τα χέρια σας παρακαλώ. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 90 είναι γλωσσική, 91 και τι ΠΕΣ 30, ΠΕΣ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. NV15 γλωσσική συμβαστική 3 Συμβαστική 3. Όχι 1 και 2. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψάρια 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Φαντάλεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 και 108 πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σαρια 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για την 110. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά αρχίζω μάλλον να κουράζομαι. Και κάτι γίνεται με το ΕΛΚ. Εψήφισαν πάντες. πέρα Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά. Σας παρακαλώ, βάλτε του, τα παιδιά να σηκώνουν τα χέρια τους. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι όμως πρέπει να ελέγξουμε. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι, γιατί οι φιλελεύθεροι πήγαν στην άλλη πλευρά. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν θα σας πω πώς τα βλέπω αυτά τα πράγματα και να σας πω τα μυστικά μου. 116 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 ή 149. 149. Το βρήκατε, 149 του κ. Φαντάλεν. Να στοιχηματίσουμε ότι αποτέλεσμα θα βγει. 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε για την 150. Νομίζω απορρίπτεται. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλά έκανα και έλεγξα. 26 πίπτη Πες 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 της εισηγητού, υπέρ, της εισηγητρίας μάλλον υπέρ, κατά, αποχές, αγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 10 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνατα. 30 ένβη προσθήκη στη συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτωτα. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωτα. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πολύ καλές σχέσεις με την Εύη αυτή τη βδομάδα ΠΕΣ 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 όχι, δεν ψηφίζουμε για αυτή. Δεν 180, 180. Grandes Πασκουάλ και Εσταρά Fragut. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 181 και 43 της Envy. μαζί, υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. 181. 181 και 43 της ΕΝΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήψαν άπαντες. Πέρασε. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. 182. Ουδίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπέρ NV44 NV44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 της αλίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. 186 έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. NV45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πες πιτς 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 και 187 μαζί υπέρ κατά αποχές να σημειώσουμε ότι εγκρίθηκε νομίζω, ε. Ωραία κύριε Βαντάλεν. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 της ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 56 της ε, ΠΕΣ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 και 189 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεκατρία. Υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλία 59. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV50. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 200 του κυρίου Κούν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201, 2 και 3 on block, προσθέτοντας ε, τους όρους με την αρμόδια υποεθνική αρχή. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υποθέτω ότι για κάποιον άλλο βγάζει νόημα. 204 του κ. Δανέλη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τι έγινε οι δύο Να ψηφίσουμε την 62 και την 63. Ωραία λοιπόν. 62 και 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και εγώ νόμιζα ότι κατέπεσε, αλλά απορρίφθηκε. Γι' αυτό έκανα αυτή την πάυση. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 207 υπέρ. 208 εγκρίθηκε. Δεν το λέει έτσι ο καταλογό μου, αλλά τέλο πάντων θα σα πιστέψω. 207 καταπίπτει. 209 αποσύρεται. 210 υπέρ κατά απόχέ Αγκρίνεται. 211 υπέρ καταπίπτει. 213 καταπίπτει, 212 αποσύρεται, 214 καταπίπτει, 215 αποσύρεται, Ναι, αλλά 206 εγκρίθηκε. Α, ψηφίζουμε το 211. Υπέρ. 211 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίβεται ούτω ή άλλω. 212 προσέχθηκε, 213 υπέρ, κατά, αποχέ, αγκρίνεται. 216. Ναι. 216 γιατί άλλες δεν εγκρίθηκαν. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία. 2.17 ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται 20 με 19 κατά. Καλά είπε ο κύριος Γκρός. Πού είμαστε τώρα? 2, όχι, 55 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.18-2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.20-2.21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 2.22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή οι επόμενες καταπίπτουν της αλίας καταπίπτει 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή αλία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 NV υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλίας 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή αλλία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλία 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Α, όχι. 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 7 της αλίας υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αλία 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αλία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλία 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται αλία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή Envy 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή NV7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή αλληλεία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ με συγχωρείτε 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άλλη 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές Ένβι NV10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλληλεία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλία 21 υπέρ κατά αποχές Ένβι NV11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αλία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μα τι σαν να είμαστε στην Επιτροπή Ελίας NV12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 της Ελίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ο κύριος Κούραν ε, μου φαίνεται ότι είναι ψαράς 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλληλεία 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 65 της αλληλείας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία κύριε και κυρία άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 32 υπέρ 7 κατά καμία αποχή εγκρίνεται τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ 7 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μάισνερ. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ρουμπίχη. Να με συγχωρείτε. Ναι. Να κάνω μία παρατήρηση, να τους ευχαριστήσω όλους ε, τους και εισηγητές ε, για την συνεργασία. Ήταν δύσκολη η έκθεση ε, γιατί ήταν κάτι το καινούριο. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολο. Η Αλία είχε μία τελείως, η Επιτροπή Αλίας είχε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Να εξηγήσω δηλαδή γιατί γίνανε έτσι τα πράγματα. Είμαι και εγώ στην Επιτροπή Αλίας βεβαίως. Σας ευχαριστώ όλους και περιμένουμε βέβαια τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ. Ασύνηθες αυτό να έχει άλλη προσέγγιση η Επιτροπή Ελίας. Έκθεση Ρούμπιχ για τα περιφερειακά σήματα ποιότητας, βέλτιστες πρακτικές της ε, οικονομίας υπαίθρου συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε νομίζω ότι απορρίπτεται άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε σας παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε την 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 34 να την επαληθεύσουμε τη 33 ωραία άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας ισοψηφία απορρίπτεται ε 34 ήταν αυτή 33 33 34 λοιπόν υπέρ κατά θα την επαληθεύσουμε γιατί δεν σηκώνει κανείς τα χέρια του. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚΑ, μάλιστα. Πέρας. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 36 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή Δύο υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται 3 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε την πέντε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Προπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, 4. Κατά καμία αποχή, συγχαρητήρια στον κύριο Ρίμπικ. yes, yes, you can. Could I ask people to leave quiet? Παρακαλώ ησυχία καθώς φεύγετε. Το επόμενο θέμα είναι η επίμαχη έκθεση για τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις για την ε, οδηγία. Η ε, σχέδιο έκθεσης, συγγετής Γιώργ Λάιχτφριντ. Κυρίες και κύριοι, Συνήθως είναι καλό να υπάρχει μία συνάντηση ε, κάθε φορά, μία συνεδρίαση. Όποιος δεν θέλει να παρακολουθεί τη συνεδρίαση, να βγει από την ε, αίθουσα. κύριε Lightfield. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήξερα ότι πρόκειται για επίμαχη έκθεση ε, μέχρι τώρα που το είπατε. Ευτυχώς που μου το είπατε για να το ξέρω Αξιότιμοι συνάδελφοι, ήταν μεγάλη μου χαρά όταν ανέλαβα αυτή την έκθεση, αφενός γιατί το θέμα είναι ενδιαφέρον, αφετέρου γιατί, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Αλλά νομίζω πως υπάρχει νομίζω ήδη μια κοινή προσέγγιση και παρακαλώ να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως κανείς εδώ πέρα δεν ήταν ικανοποιημένος από το πώς είχαν κυλήσει τα πράγματα και νομίζω πως ε, είχαμε ένα καλό παράδειγμα του πώς δεν πρέπει να προετοιμάζονται οι νόμοι. Επειδή όμως το έχω πολλές φορές δεν θα το επαναλάβω τώρα. Για την ίδια την έκθεση θεωρώ πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον νομοθέτημα το οποίο βεβαίως ε, έχει κάποια στοιχεία με τα οποία διαφωνώ. Εγώ θεωρώ πως είναι προς το κοινό συμφέρον μας ε, η οδική κυκλοφορία να γίνει πιο οικολογική, να μην βλέπουμε τη διάφορα μέσα μεταφοράς ως ε, εισάξια, αλλά κάποια να θεωρούμε πως πρέπει να ενισχυθούν περισσότερα. 8,5 χρόνια ακολούθησα αυτή τη γραμμή, μέχρι πριν από λίγους μήνες, όταν υπήρξαν κάποιες τάσεις που εγώ τις θεωρώ λανθασμένες. Αυτή η κοινή λογική, δηλαδή να λέμε πως ε, θέλουμε να υπάρξει μια μετατόπιση από τους δρόμους στο σιδηρόδρομο, ε, θεωρώ πως ε, πλέον είναι κάτι το οποίο δεν τηρεί η Κομισιόν και ο Επίτροπος Κάλλας. Αντιθέτως, θεωρώ πως πάει σε μία διάσπαση αυτής της ε, συνένεσης. Είναι λανθασμένο, λανθασμένη αυτή η προσέγγιση, δεν είναι αυτή η πολιτική που χρειάζεται η Ευρώπη, είναι η πολιτική που χρειάζονται κάποιοι λομπίστες ε, και είναι ε, προς το συμφέρον κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων και όχι υπέρ του γενικού συμφέροντος. Οπότε έκανα κάτι το οποίο σπάνια έχω κάνει, δηλαδή επί της αρχής απέρριψα την πρόταση της Κομισιόν και ε, άλλαξα τελείως το, το νόημα και το περιεχόμενό της. Αυτά τα οποία δεν λέει η Κομισιόν, τα μισόλογα με τα οποία προσπαθεί να περάσει το ότι θέλει να επιτρέψει τα πολύ μεγάλα φορτηγά να περνάνε τα σύνορα είναι κάτι το οποίο πλέον αλλάζει την πορεία δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι λόγοι είναι προφανείς. Εάν δει κανείς την πρόταση της Κομισιόν και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ συνάδελφοι διαβάζει κατά λέξη το εξή. Ε, ήταν μέχρι τώρα έτσι η κατάσταση, ήρθαν κάποιοι ενδιαφερόμενοι στον ε, Επίτροπο, οπωσδήποτε δεν θα ήταν πρόσκοποι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι και έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση προς το συμφέρον ε, των εταιριών των μεταφορών. Έτσι ξεκίνησε η όλη υπόθεση. Και θα δούμε τι θα προκύψει. Εγώ πρότεινα στο μέλλον να μην επιτρέπονται διασυνοριακά ταξίδια αυτών των μεγάλων ε, φορτηγών ε, στην Ευρώπη στο μέλλον. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό το οποίο υπήρχε στο κείμενο, δηλαδή κάποιες γενικότητες για την ασφάλεια, κάποιες γενικότητες για την καλύτερη επιτήρηση του βάρους, να συνδεθούν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα είναι βεβαίως ε, παρκές για προετοιμασία αλλά να πάμε σε κάποιες ε, δεσμευτικές ε, διατάξεις και είναι σημαντικό νομίζω να δούμε και την ασφάλεια των υπολείπων που βρίσκονται στον δρόμο. Και πρέπει άρα οι μηχανισμοί αυτή προστασίας να είναι υποχρεωτικοί. Επίσης θεωρώ πως στο μέλλον θα πρέπει να είναι η δυνατότητα να ελέγχουμε καλύτερα το βάρος και γρηγορότερα, ειδικά οι αρχές που έχουν μεγάλες δυσκολίες και απαιτούνται πάρα πολύ πόροι για αυτή τη δουλειά. Και ακριβώς εδώ πέρα είναι το θέμα το εάν στέκει επιστημονικά ή όχι κάτι τέτοιο. Εγώ έχω νομίζω μαζέψει αποδείξεις για το ότι στέκει και θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικές ενδείξεις του βάρους στο μέλλον τα φορτηγά για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και για να προστατεύουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς που δεν μπορούν να εκτιμήσουν πόσο βαριά φορτωμένο είναι ένα φορτηγό. Για το θέμα των αεροδυναμικών μέτρων, επί της αρχής είμαι θετικός. Βεβαίω υπάρχει ήδη μια οδηγία η οποία καθορίζει ποια μέτρα επιτρέπεται να ληφθούν, πόσο μεγάλες μπορεί να είναι αυτές οι συσκευές. Η πρόταση της ε, Κομισιόν είναι αντίθετη με αυτή την οδηγία, η οποία συμπτωματικά βεβαίως είναι μιας άλλης γενικής διεύθυνσης. Και προσπάθησα και εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να είναι στο μέλλον υπό είναι συμβατά στο μέλλον. Θετικό είναι επίσης οτιδήποτε συνεισφέρει στην ε, μικρότερη κατανάλωση μεζίνης ε, καυσίμου από τα συνηθισμένα φορτηγά. Αλλά και εδώ πέρα προσπαθήσαμε να μείνουμε ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία. Να επιτρέψουμε δηλαδή και άλλους ε, τρόπους ε, κίνησης ε, των φορτηγών, έστω και αν γίνονται έτσι βαρύτερα τα φορτηγά, κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως βεβαίως δεν μας δίνει την εντύπωση πως θα είναι πιο οικονομικά στην κατανάλωση καυσίμου. Αυτό λοιπόν το οποίο σας παρουσίασα αγαπητοί συνάδελφοι είναι η δική μου η πρόταση. Ξέρω πως ειδικά οι σκιώδεις εισηγητές βλέπουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Ξέρω επίσης πως τελικά θα πρέπει να βρούμε έναν συμβιβασμό τον οποίο θα στηρίξει η πλειοψηφία για να έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα για την Ευρώπη. Καλό για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για όσους μένουν κοντά σε οδικούς άξονες και για τους φορολογούμενους. Δεν είναι νομίζω σωστό να αλλάζουμε κάποια πράγματα και να πληρώνει κάποιος την υποδομή την οποία θα χρησιμοποιούν ε, άλλοι για να βγάλουν κέρδος. Ήμουν και σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου ένας εκπρόσωπος ενός κράτους μέλους που τα βλέπει θετικά αυτά τα θέματα και θεωρεί πως Συνολικά το κόστος για την επιδιόρθωση των δρόμων είναι 40 εκατομμύρια ευρώ και το κέρδος των επιχειρήσεων είναι ε, πολύ μεγαλύτερο. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα νομίζω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους ε, σκιοδησίτες παρά το ότι κάπου αποκλίνουν οι ιδέες μας για την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία μας. Και πρέπει να αναγνωρίσω πως ε, οι υπόλοιπες προτάσεις, οι οποίες δεν ανέφερα ακόμα, είναι νομίζω λογικές και θεωρώ πως τελικά είμαστε σε θέση να βρούμε μια συμβαστική λύση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λόγκφριντ από την Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική για τρία λεπτά ο κύριος Ρίνο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ήμουν ο, ο εισηγητής της ΕΚΟΣΟΚ για αυτήν την πρόταση για τις διαστάσεις και το βάρος. Το έγγραφο, η γνωμοδότησή μας, συζητήθηκε κατά την Ολομέλεια του Ιουλίου και εγκρίθηκε ομόφωνα, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντοτε. Διαβάζοντας τώρα το σχέδιο έκθεσης το δικό σας, βρίσκω ότι πολλά σχόλια και προτάσεις ε, εναρμονίζονται με ό,τι προσπαθήσαμε να πούμε και εμείς στη δική μας έκθεση. Μεταξύ άλλων ένα παράδειγμα, όταν βλέπουμε το πλεόνασμα βάρους, ο κύριος Λάιτφιλτ με τις τροπολογίες του αναφέρει τον όρο ε, οχήματα εναλλακτικής τεχνολογίας για να επιτύχει αυτή την τεχνολογική ουδετερότητα την οποία και εμείς στηρίζουμε. Εν τέλει όμως, δεν ξέρουμε πόσο καλή θα είναι η οδηγία. Παρά μόνο μετά από την υιοθέτηση των πράξεων κατ' θα το μάθουμε. Ασφαλώς το ξέρετε αυτό. Και σίγουρα θα συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε το θέμα. Χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, επιτρέψτε μου να θίξω έτσι μερικά θέματα για να συμβάλλω κι εγώ στην συζήτηση. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να προσφέρω, γιατί δεν το είδα στη δική σας έκθεση, έχει να κάνει με το άρθρο 16β της πρότασης, το οποίο μιλά για μονάδες ε, μέγιστου μήκους 40 με 45 ποδιών μέχρι 44, μέχρι 44 τόνους για, για οχήματα τριών αξώνων. Κατά τη γνώμη μας η πρόταση αυτή θα πρέπει να ισχύσει και για τα οχήματα με δύο άξονες. Θα θυμάστε ότι πάνω από το 90% των κυκλοφορούν των οχημάτων στην Ευρώπη έχουν δύο άξονες. Το να περιορίσουμε τη ρύθμιση αυτή στα οχήματα με τρεις άξονες δεν θα βοηθήσει την κατανάλωση αλλά και ακόμα πιο σημαντικό, δεν θα ωφελήσει τις ενοποιημένες μεταφορές για την αντικατάσταση του κυκλοφορούντος τόλου οχημάτων. Μετά, έχουμε ε, αυτά τα μέγα φορτηγά, τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Τώρα για τα υπέρ και τα κατά του EMS, τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά, καταλαβαίνω ότι πολλοί μεταξύ των οποίων και ο εισηγητής, θεωρούν τα, επί, τα σκέφτονται ε, να, υπάρχει ένα, να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα. Εάν έχουμε αυτή τη διασυνοριακή χρήση των VMS, υπάρχει η πιθανότητα να επέλθει ένα φαινόμενο ντόμινο ε, για τα οχήματα σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα ενδεχόμενο. Εάν συμβεί αυτό, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν θα μπορεί παρά να σημειώσει το γεγονός και θα αφήσει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν εκείνα πώς θα συνεχίσουν. Εάν τα μακρύτερα οχήματα κερδίσουν ένα μερίδιο αγορά. σε εκείνα τα κράτη-μέλη όπου υπάρχει κατάλληλη υποδομή και εξασφαλίζονται οι όροι ασφάλεια στο εσωτερικό τους δίκτυο, δεν είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει τα κράτη αυτά χωρίς να παραβιάσει την αρχή της επικουρικότητας, την οποία διεκδικούμε κάθε λίγο και λιγάκι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είχα και άλλα σχόλια, αλλά επειδή βλέπω ότι δεν έχω άλλο χρόνο, θα σταματήσω εδώ και θα ξαναευχαριστήσω τον Πρόεδρο και όλους εσάς για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχω και πολύ μεγάλο κατάλογο ομιλητών, όπως ε, θα φαντάζεσαι. Μάλλον έχω ένα μακρύ κατάλογο ομιλήτων, όπως θα φαντάζεσαι και θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ όπως κάνω συνήθως. Τρία λεπτά για τους κεώδεις εισηγητές και δύο λεπτά για τους υπόλοιπους ε, ομιλητές. Έχω τους σκιώδεις εισηγητές και μετά μια σειρά ομιλητών, 5 με 6 με τελευταίο τον κύριο Μπαχ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος και για άλλους, αλλά αν θέλει και κάποιος άλλος να προσθεθεί, ο κύριος Γκρός, μάλιστα. Ε, βάζω το ρολόι με τον κύριο μου ο καθένας θα έχει τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Εισηγητή για τη δουλειά σας. Καταρχήν θα κάνω ένα σχόλιο εδώ. Εσείς κύριε Λάιτφριντ χρησιμοποίησατε το 80 με 85% του χρόνου σας για, τις, για την διασυνοριακή κυκλοφορία των μακρών οχημάτων. Αυτό νομίζω κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Δείχνει σε όλους ότι ε, αυτή είναι η ουσία του ζητήματος, ότι αυτό είναι το θέμα. Παρόλο που στην αρχή δεν ήταν αυτή η πρόθεση και υπήρχαν πολλά καλά επιχειρήματα και πολύ καλές ρυθμίσεις για την αποδοτική χρήση των καυσίμων, για τα βάρη, για, την αεροδυνα... για τις αεροδυναμικές προδιαγραφές. Ασφαλώς όλα αυτά τα χρειαζόμαστε και αυτά είναι πολύ σημαντικά στην πρόταση αυτή της Κομισιόν. Επιτρέψτε μου όμως και εγώ να αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής μου στη διασυνοριακή κυκλοφορία των οχημάτων. Ξέρουμε ότι η μεταφορά αγαθών θα αυξηθεί στο μέλλον και μάλιστα πάρα πολύ. Θα φτάσει γιγαντιές διαστάσεις. Ξέρουμε ότι στις χώρες όπου χρησιμοποιούν αυτά τα ελαφρώς μεγαλύτερα φορτηγά με τους ε, με τα διαφορετικά αξονικά γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στις χώρες εκείνες που χρησιμοποιούν επί πολλά χρόνια αυτά τα οχήματα, σε μερικές χώρες για 15 χρόνια. Ξέρουμε και ότι υπάρχουν ουσιώδη οικονομικά πλεονεκτήματα. Ε, και ξέρουμε ε, ότι ξέρουμε σίγουρα ότι δεν τίθενται θέματα ασφάλειας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει για τα ευρωπαϊκά κράτη που χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο των 30-35 μέτρων. Και ακόμα πιο σημαντικό, γνωρίζουμε σίγουρα ότι στις χώρες αυτές το μερίδιο των σιδηροδρόμων, ένα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας εδώ, είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Στην Φιλανδία είναι 25%, στη Σουηδία, στη Δανία. Αυτό που είναι ακατανόητο για μένα είναι το εξή. Όταν όλα τα στοιχεία και όλα τα γεγονότα που έχουμε δείχνουν μια ελεύθερη κυκλοφορία, έτσι ώστε να, μπορέσουμε, να αντικαταστήσουμε τα φορτηγά στο δρόμο. Όσο λιγότερα φορτηγά υπάρχουν, τόσο λιγότερα ατυχήματα γίνονται, τόσο λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπεται και ακόμα πιο σημαντικό ίσως, μοιάζει να μην υπάρχει μια μετάβαση από το σιδηρόδρομους στους δρόμους λόγω αυτών των οχημάτων, ε, μου δημιουργείται μια μηχανία και θα με καταλάβετε που εκφράζω αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Σοβάνα. Κάποιοι, συμφωνούν εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, ενθουσιοδός. Ε, Κύριος Μπένιαν, για τους φιλελεύθερους. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του πάνω στην έκθεση αυτή. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ασφάλεια και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα φορτηγά. Και θα ήταν κρίμα να μην επιτύχουμε την πρώτη ανάγνωση. Η προθεσμία για τις, ε, η καθυστέρηση της, ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ελπίζω ότι δεν θα καθυστερήσει περαιτέρω την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις για τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις ε, στην εθνική και διεθνή κυκλοφορία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν οι γεωγραφικές πραγματικότητες. Γενικά δεν είμαι υπέρ των πιο βαρέων οχημάτων και των μεγαλύτερων οχημάτων γιατί υπάρχει μια κοστοβόρα υποδομή από πίσω. Όμως, ε, εδώ ανακύπτει και ένα άλλο ζήτημα που είναι το ύψος των οχημάτων. Ο εισηγητής, ε, όταν κατέθεσε την έκθεσή του, δεν ξέρω αν έλεβε υπόψη του τα όρια ύψου στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πολύ υψηλά οχήματα που κυκλοφορούν μεταξύ Ιρλανδία και Ηνωμένου Βασιλείου για πολλά χρόνια και θέλουμε να, να, σταματήσουμε αυτά τα άνω των 4 μέτρων ε, οχήματα να, να πηγαίνουν στην Βόρειο Ιρλανδία. Επίσης πρέπει να βρούμε μια λύση που να ε, αντιμετωπίζει την περίπλοκη πραγματικότητα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Σε μερικά κράτη-μέλη που υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν τα θέματα στα σύνορα και υπάρχουν και τα θέματα της ενιαίας αγοράς. Για τις, ε, για το, για τις αεροδυναμικές προδιαγραφές είμαι με το μέρος του εισηγητή. Γενικά είμαι υπέρ, αλλά μοιάζει να υπάρχουν κάποια προβλήματα με την υφιστάμενη νομοθεσία και τις διαδικασίες έγκρισης. Θα ήθελα η Κομισιόν να το διευκρινίσει αυτό. Τώρα, πάλι υπερ... είμαι με τον εισηγητή όσο αφορά τις βελτιώσεις που μπορούμε να υποφέρουμε, αλλά θέλω να δώσουμε και τον κατάλληλο χρόνο στους κατασκευαστές. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες για τα αστικά φορτηγά, όπου εκεί η αεροδυναμική δεν παίζει και τόσο σημασία. Τώρα, οι συνδυασμένες μεταφορές, οι συνδυασμένες εξαγωγές, δυστυχώς καθώς όπως έχει ο ορισμός αυτήν τη στιγμή, πολύ φοβάμαι ότι εξαιρούνται κάποια οχήματα από, την, τον σημερινό ορισμό των συνδυασμένων μεταφορών. Ή θα πρέπει να αλλάξουμε τον ορισμό ή κάτι άλλα μέτρα, κάποια άλλα μέτρα να λάβουμε. Νομίζω ότι συμφωνώ ότι δεν μπορούν να υπάρχουν συνδυασμένες μεταφορές με τεράστια, μεταξύ τεράστιων ταξιδιών και μικρών ταξιδιών ή διαδρομών. για τα χιλιόμετρα τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό με την Κομισιόν, γιατί πρέπει να είμαστε αυστηροί. Ο κύριος Γκράμερ για τους Πρασίνους για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συγητή, ειδικά για τα ξεκάθαρα λόγια που είπε στην αρχή. Εμείς καταφέραμε να μην παραβιάσει το δίκαιο εδώ πέρα ο Επίτροπος. Γιατί ε, δεν ήθελε να αλλάξει τον νόμο, ήθελε να κάνει μια διαφορετική ερμηνεία. Δεν είναι αυτό το πράγμα λειτουργία κράτους δικαίου. Ανεξαρτήτως τις θέσεις που έχει κανεί εδώ πέρα στην Επιτροπή, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ότι δεν το ανεκτήκαμε. Δεύτερον, οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά θετικά στην έκθεση, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. 50% της, της συνδυασμένης μεταφοράς στην Ευρώπη πήγε, μεταφέρθηκε στις, ε, στους, στους δρόμους. Δεν μπορεί να εξοικονομηθεί, λοιπόν, να εξοικονομηθούν όλες αυτές οι εκπομπές ε, με τα Megatrax. Οπότε το 20% μείωση που είχαμε αποφασίσει μέχρι το 2020 στην έκθεση Ματιά Γερός πρέπει να ενσωματευτεί. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το τρίτο και το τέταρτο βήμα χωρίς το πρώτο. Και άλλα θετικά σημεία είναι σκαμπίνες ασφαλείας. μα το σχέδιο μετά τη μεταβατική περίοδο πρέπει να είναι ε, δεσμευτικό. Ε, η Κομισιόν Μα μας έλεγε άλλα πράγματα. Εδώ πέρα το βάλατε πράγματι θετικό στην έκθεσή σας. Διασυνοριακές μεταφορές πρέπει πράγματι να μειωθούν και αυτό είναι θετικό στην έκθεσή σα, Εναλλακτικά καύσιμα, σωστό. Τεχνολογική ουδετερότητα, δεν είμαστε μηχανικοί εμείς. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να λέμε πώ θα επιτευχθεί και επίση και η προστασία των πεζών σημαντική πού μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση. Δυνατότητες ελέγχου τήρησης όλων αυτών των πραγμάτων. Πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρός ο έλεγχος. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα της Κομισιόν. Γράφει εδώ πέρα νέους νόμους, αλλά δεν φροντίζει το να τηρούνται. Ε, νόμοι που δεν τηρούνται δεν χρειάζεται να τους γράφουμε καν. Έτσι. Γλιτώνουμε και τον κόπο μας. Απευθύνω έκκληση λοιπόν στην Κομισιόν να τηρηθεί η υπάρξη νομοθεσία. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα, όχι να γράφουμε κάθε εβδομάδα νέους ε, νόμους. Ε, τα Gigaliner καλύπτονται εδώ πέρα. Όπως είπα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους 20% και υποδομές. Ε, προσπεράσεις, ε, το πώς καθυστερεί η κυκλοφορία, η κατασκευή νέων δρόμων. Ήδη η Αυστρία θα πρέπει να δώσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών. Και ε, τι έχουμε εδώ πέρα, κοινωνικοποίηση της χασούρας και ιδιωτικοποίηση των κερδών. Θα ήμασταν χαζοί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό στηρίζουμε την έκθεση του εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Φαντάλεν για τρία λεπτά. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς ε, τους ε, συναδέλφους για την καλή συνεργασία. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο ένα πρόβλημα υπάρχει εδώ πέρα. Ε, πάτε σε τελείως λάθο κατεύθυνση. Ε, συμβαίνουν αυτά σοσιαλιστέ. αλλά εδώ πέρα είναι πολύ, δηλαδή τα πράγματα είναι ιδιαίτερω άσχημα. Ναι κύριε Πρόεδρε. Α δούμε δηλαδή μόνο την ορολογία. Μιλάτε για monster trucks και τέτοια πράγματα. Όχι, είναι οικολογικά φορτηγά. Είναι καλά για το περιβάλλον. Γιατί μειώνουν με το να είναι μεγαλύτερα σε μήκο και την κατανάλωση και την επιβάλληση του περιβάλλοντος. Καλό είναι να τα λέτε λοιπόν οικολογικά ή οικονομικά φορτηγά. Και βεβαίω κλασική περίπτωση έχετε μια λογική προσανατολισμένη προς ε, το κράτος το οποίο θα επιβάλλει περιορισμού κτλ. Και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και τα πειράματα έχουν αποδείξει πως ε, και στον τομέα της ασφάλειας, της εκπαίδευση των οδηγών, ε, όλοι οι χρήστε αυτών των φορτηγών λένε ναι, αυτά είναι πραγματική βελτίωση. Και ο, ο... με ο εδώ πέρα έρχεται και λέει όχι, όχι, δεν τα θέλουμε, δεν θέλουμε βελτίωση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς του εισηγητή μας. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να συμφωνήσω εδώ πέρα καθόλου και το είπε και ο εισηγητής των χριστιανοδημοκρατών. Η κίνηση θα αυξηθεί. Έχουμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ καλό μέσο το οποίο μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε την αύξηση της κίνησης με τρόπο ασφαλέστερο και φιλικό προς το περιβάλλον. Ε, δηλαδή είναι κατόρθωμα να είναι κανείς εναντίον. Ε, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι κανείς κατά. Εντάξει, εμείς μπορεί να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Ε, γιατί ήταν και σύντομες ούτως ή άλλως και οι συναντήσεις των συντονιστών γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι διαφωνούσαμε και μπορούμε απλά δηλαδή να λέμε υπέρ ή κατά ή οικολογικά φορτηγά ή master tracks όπως τα λέει ο καθένας και να τελειώσει εκεί η υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ησυχία. Λοιπόν, ο κύριος Ήκε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Είμαι με το μέρος του εισηγητή, παρόλο που το ΕΛΚ ε, δεν είναι πάντοτε με το μέρος του. Υπάρχουν δύο μέρη. Υπήρχαν αυτοί που είναι υπέρ των μεγάλων ε, φορτηγών, εκείνοι που είναι κατά των μεγάλων φορτηγών. Ε, όλοι έχουν κατανοήσει ότι οι επιδόσεις των χερσαίων, ε, στις χερσαίες μεταφορές οι επιδόσεις των μεγάλων φορτηγών είναι καλύτερες και αν υπάρξει η κατάλληλη υποδομή θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις, ακόμα καλύτερες επιδόσεις, θα μεταφέρονται περισσότερα αγαθά κτλ. κτλ. Βέβαια το γενικό κοινό δεν είναι ευχαριστημένο με αυτά τα τερατώδη οχήματα γιατί υπάρχει αυτή η ανισότητα. Υπάρχει το οδικό δίκτυο το κατάλληλο για τα μεγάλα φορτηγά και υπάρχει και το οδικό δίκτυο που είναι κατάλληλο για τα υπόλοιπα οχήματα. Και πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε τα συμφέροντα όλων των οδηγών φορτηγών. Αν ε, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αν βάλουμε περισσότερα μεγάλα οχήματα στους δρόμους και μεταφέρονται περισσότερα αγαθά, σίγουρα θα μειωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Αν το δείτε όμως μακροπρόθεσμα, εάν μεγαλώσει ο στόλος και κυκλοφορούν περισσότερα οχήματα, τότε φυσικά οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα θα είναι πολύ περισσότερες εν τέλει. Ε, και πάντως αυτά που ισχύουν για τα μεγάλα φορτηγά δεν μπορούν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν παντού στην Ευρώπη. Ε, δηλαδή υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Ε, εσείς μιλάτε για το μεσαίωνα τώρα. Ε, ναι, κάποια πράγματα, ορισμένα κομμάτια της υποδομής θυμίζουν το μεσαίωνα. Δεν είναι δυνατόν να εξυγχρονιστούν εν μία νυχτή. Πρόεδρος. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο ησυχία. Κύριο Σερτούγ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Σπάνια συμφωνώ τόσο απολύτως όπως σε αυτή την ε, περίπτωση. Δεν είναι έκπληξη. Θα αναφερθώ στα βασικά επιχειρήματα στα δύο αυτά λεπτά. Πρώτον, ε, ξεκάθαρα θα πρέπει να πάμε σε μια μετατόμιση της ε, κυκλοφορίας σε πιο ε, φιλικές μορφές μεταφορών. Υπάρχει μια μελέτη που τα αποδεικνύει αυτά και δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής καμία αντίρρηση που να είναι υπέρ της αγωγής των Gigaliner. Έχουμε τις εξελίξεις Σκανδιναβία και στις κατοχώρες όπου είχαμε ξεκίσει με μια σαλαμοποίηση με τους 40 τόνους, εντωμεταξύ έχουν περάσει τους 60 τόνους και πάνω. Μιλάω για το βάρος των φορτηγών. Αυτό το οποίο θα ήθελα να υπενθυμίσω είναι πως ε, πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε και μια συνεπή πολιτική έτσι και εδώ πέρα μιλάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν από τη μία να λέμε λευκή βίβλος ε, ε, για την κυκλοφορία και να ορίζουμε πώς θα πρέπει να μεταφερθεί η κυκλοφορία στους σιδηρόδρομους και μετά να φέρνουμε αυτή την νομοθεσία. Δεν υπάρχει επίσης εδώ πέρα αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν που θα αποδεικνύει αυτά τα οποία λέει. Έτσι. Και να πω κάτι άλλο όσον αφορά το κόστος της υποδομής. Και πραγματικά ε, είναι αντικείμενο και των διαπραγματεύσεων στη Γερμανία για το σχηματισμό κυβέρνησης και έχουν κολλήσει στα διόδια για τα ΙΟΤΑΧΗ, έτσι, τα οποία θα εισαχθούν για πρώτη φορά στην ε, Γερμανία για να μπουν λεφτά στα ταμεία και με αυτά που ακούω, τι να πω, ε, ας ξεκινήσουμε καλύτερα από τα μεγάλα, έτσι, τα, τα διόδια για τα φορτηγά, να τα προσαρμόσουμε πραγματικά για να πληρώνουν περισσότερα και μετά να επεκταθούμε και στους αυτοκινητόδρομους και στην εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Ε, Βεβαίω εσείς μας μιλάτε για το επιχειρηματικό συμφέρον γιατί αυτά σας λένε τα λόμπι. Ε, εντάξει, κατανοητό να ε, γίνουν τα περισσότερα φορτηγά λιγότερα, αλλά το κόστος θα γίνει μεγαλύτερο για τις ε, υποδομές. Και να σου πω κάτι άλλο, οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που θα υποφάρουν, γι' αυτό, γι αυτό ακριβώς είναι κατά των τεράστιων αυτών φορτηγών. Κύριε Ντεμπάκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για αυτά τα οποία είπε. Πράγματι θετικά αυτά τα οποία μίλησε για την ε, αεροδυναμική και τα λοιπά, θετικά αυτά, αλλά σήμερα συζητάμε κάτι άλλο. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, ανατρέπει τελείως την πολιτική των μεταφορών. Και τι θέλει να μετατοπίσει τις μεταφορές ξανά από το σιδηρόδρομο στο δρόμο. Νόμιζα πως πηγαίναμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κοιτάξτε όμως ο σκοπός μας εδώ πέρα δεν είναι το θέμα να βάζουμε εμεί εμπόδια. Αν υπάρχει κάποια καινοτομία που κάνει καλύτερη τη μεταφορά στους ο, δρόμους πρέπει και ο εισηγητής εδώ πέρα να μην βάζει εμπόδια και να ανατρέπει την ε, πολιτική, την υφιστάμενη. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, ο εισηγητής βάζει ξανά εμπόδια στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οδικών μεταφορών. Ε, κάτι το ασύλληπτο. Κάτι άλλο επίσης που δεν αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μεταξύ Γαλλίας ε, και χωρών Μπενελούξ για τα φορτηγά των 54 ε, τόνων. Εκεί πέρα είναι το, το όριο. Νομίζω πως θα πρέπει να επικρατήσει λογική και να βρεθεί μια συνεννόηση μεταξύ των ε, χωρών. Συμπέρασμα. Όποιος θέλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πιο ευρωπαϊκή και πιο ολοκληρωμένη πολιτική μεταφορών θα πρέπει να υποστηρίξει την καινοτομία και να αφαιρέσει τα εμπόδια που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ κυρία Φώστερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ να συμφωνήσω με μερικά από τα μερικές από του κυρίου Φαντάλεν. Πρέπει βεβαίω να μην ξεχνάμε και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και έχω ζήσει και στην Αυστρία. Ξέρω τι γίνεται εκεί με τα σταυροδρόμια και καταλαβαίνω και τι δικέ του ανησυχίε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να δούμε και την πρόοδο τη τεχνολογία, τι γίνεται με τα φορτηγά και το τι γινόταν πριν από μία δεκαετία. Είναι τεράστια η εξέλιξη. Ε, Κάποιε φορέ δεν τα λαμβάνουμε παρκώ υπόψη. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Οι αποστάσει από, από γεωγραφική άποψη δεν υπάρχουν συνδυοδρομικέ ανταποκρίσει. Πρέπει λοιπόν τα φορτηγά να διανύσουν τεράστιε αποστάσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι φτάνουν στο κέντρο τη πόλη. Πολλέ φορέ τα αγαθά ε, μεταφέρονται σε μια αποθήκη και μετά φτάνουν στο κέντρο τη της Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Από την άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θέλουμε τίποτα να διακυβεύσει, την, ε, να, να θέσει σε αμφιβόλο την ε, οδική ασφάλεια. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν όλες τις σχετικές τροπολογίες. Για τα α, οχήματα τα οποία κινούνται με αέριο, θα, με βενζίνη μάλλον θα το... Θα δεχτούμε κάθε σχετική εξέλιξη, αλλά για την ώρα έχουμε τα φορτηγά των 4 μέτρων, τα οποία κυκλοφορούν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, και δεν βλέπουμε το λόγο να αλλάξει κάτι σε αυτή την παράδοση. Ω προ την αόριστη περίοδο για τι καταξιοδότηση πράξεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν το στηρίζουμε αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε πάλι να τα ξανασκεφτόμαστε. Αλλά για κάποια από τα άλλα πράγματα που υπόθηκαν. Καταλαβαίνω το σημείο αφετηρία του συγκεκριτή, αλλά θα πρέπει να δώσουμε κάποιο νόημα στην όλη συζήτηση και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια εύστοχη πρόταση. Δεν θέλουμε εμεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επιβάλλουμε στι υπόλοιπε χώρε τι θα κάνουν. Όχι. Να υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασία. Αλλά αφού θέλουμε διασυνοριακή συμφωνία και διασυνοριακέ παραχωρήσει, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με ρεαλιστικό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι μέρημνε έχουμε η ΜΕΝ και η ΔΕ, τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβουμε σοβαρά υπόψη τι προτάσει που έχουν γίνει. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο λογικό συμπέρασμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω τώρα. Ο κύριο Ρικέ θα αναλάβει. Μάλλον ο κύριο Βαντάλεν. Αλλά επόμενη μιλήτρια, κυρία Βορτμαν Κόλ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω τα σχόλια του κυρίου του κυρίου Φαντάλεν και τη κυρία Φώστερ το πρώτο πρόβλημα στη συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου, είναι ότι υπάρχει πολύ συναισθηματισμό. Δεν βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα αρκετά. Ο κ. Λάιχτφριντ μίλησε για τι ομάδε άσκηση πίεση. Ναι, υπάρχουν ασκήσει ε, πίεση υπέρ, αλλά και κατά από το σιδηροδρομικό χώρο, λόγω χάρη στι κάτω χώρε. Έχουμε κάποια hot spot ε, λογιστική μέρημνα ε, που δεν υπάρχουν ανταποκρίσει και εκεί τα βαρέα οχήματα ε, εξασφαλίζουν τις μεταφορές και είναι αποτελεσματικότερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο ούτε οικολογικά φορτηγά, ούτε gigaliner, ε, τα μέγα φορτηγά. Η εμπειρία μας από τις κάτω χώρες είναι ότι δεν χρειάζεται περιττέρω κόστος για τις υποδομές, διότι οι αποστάσεις υπολογίζονται μόνο για ορισμένα φορτηγά. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας, διότι αυτοί οι οδηγοί ουσιαστικά έχουν επιπλέον κατάρτιση. Υπάρχουν λοιπόν πρόσθετα εχέγγυα στο όλο σύστημα και είναι κάτι που δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο ούτε επίμαχο στις κάτω χώρε. Για ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και δεν καταλαβαίνω το εξής. Ζούμε σε μια ενιαία Ευρώπη. Αυτό προτείνει ο συγκεκριτής. Είναι Εάν προτείνουμε και δεχτούμε κάποια φορτηγά στι κατοχώρε, στα σύνορα του Βελγίου και τη Γερμανία, λόγω χάρη, να επιτρέπονται και στο Βέλγιο. Και τα κοντινά κρατήρια τη ε, Γερμανία, η Βεσταλία να, να τα επιτρέψει. Μιλάμε για τη συνοριακή Ευρώπη. Θα ήταν γελίο να μην γίνεται αυτό. Άρα, εγώ θα ήμουν υπέρ του να υπάρξει ένα σύστημα αδειοδότηση στα κράτη-μέλη που να ισχύει για ορισμένα μόνο φορτηγά μεν, αλλά να μην απαγορεύουμε τα σαφάτα φορτηγά να περάσουν τα σύνορα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το ότι τηρήσατε και το χρόνο. Ο Μπράιαν είπαμε πως θεωρεί θετική αυτή η πρόταση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Higgins, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με τα σχόλια. της ε, Πέτρα, του τον Ιμπάνιαν, ε, τα δικά σας κύριε Φαντάλεν και άλλων συναδελφών. Είναι γελίο το θέμα. Εντάξει, ξέρω πως έχει ως αφετηρία το περιβάλλον, αλλά αν δείτε την κατάσταση. Τα, τα μεγαλύτερα φορτηγά σημαίνει λιγότερος, μικρότερος αριθμός φορτηγών. Έτσι. Και λιγότερη οδηγή και μικρότερο κόστος. Αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, πως κατά την άποψη σας είναι απαράδεκτο αυτό. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω Ιρλανδικά και δεν ζητάω συγγνώμη. Εμείς είμαστε νησί, δεν έχουμε αποστάσεις για να αναπτύξουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς ε, έχουμε μία υποδομή ε, στο μέτρο των 4,65 μέτρων. Γιατί λοιπόν εμείς να τιμωρηθούμε για την υποδομή μας, ε, για να επιτρέψουμε ψηλότερα και μεγαλύτερα φορτηγά. 95% του στόλου μας είναι πάνω από τα 4 μέτρα, εξάγουμε, εξαρτώμεθα και από τα ferry boat, τα οποία επίσης είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Εξηγώ, εξηγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν το πόσο ωφελείται εδώ πέρα ο κλάδος, το διασυνοριακό εμπόριο και σε γενικές γραμμές είναι λογική νομοθεσία. Όμως ποτέ δεν θα υπερασπιστώ, δεν θα δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα. Τροπολογία 16 είναι αδικαιολόγητη. Είναι κατά των επιχειρήσεων και μιλάτε για σιδηρόδρομο. Δεν υπάρχει σιδηρόδρομο στη χώρα μου. Δεν έχουμε τέτοια υποδομή. Οπότε θα είμαι ιδιαίτερος κατά αυτού του μέτρου. Και από περιβαλλοντική και οικονομική και οποιαδήποτε άλλη σκοπιά. Σας ευχαριστούμε κύριε Higgins για το ότι ρίσατε το χρόνο. Μπαχ. Η κυρία Μπαχ, ο κύριος σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα βλέπουμε την ποικιλομορφία της Ευρώπης. Έχουμε αλπικές περιοχές, χώρες διέλευσης, νησιωτικά κράτη. Γι' αυτό και δεν ζηλεύω τη θέση του εισηγητή, που κατά την άποψή μου υπέβαλε μια καλή έκθεση, αλλά δεν ζηλεύω και τους κοιόδης εισηγητές. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, ο συνάδελφος του ΕΛΚ ε, είναι σε, δύσκολη θέση. Εγώ δεν θα μπω στο θέμα ε, συναισθηματικά. Το θέμα βεβαίως ε, είναι το κόστος. Ε, το κόστος όμως αυτή τη στιγμή και ο υπολογισμός του κόστους δεν βασίζεται σε επιστημονικά νούμερα. Τα νούμερα είναι ανάλογα με το λόμπι του καθενός. Καμιά φορά είναι και γελία κιόλας. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να μπω τώρα στη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια ουσιαστική μελέτη αντικτύπων για να έχουμε αξιόπιστα νούμερα. Όσον αφορά τη μετατόπιση από το σιδηρόδρομο στο δρόμο, μείωση εκπομπών, κόστος της υποδομές, η πλευρά της ασφάλειας, όλα αυτά ε, νομίζω πως δεν παρουσιάζονται ικανοποιητικά για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ντεμπάκερ ε, δεν έχουμε πει τίποτα για τους 44 ε, τόνους, οπότε εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω στη συζήτηση. Μάλιστα, σας ευχαριστώ που τηρήσατε και εσείς τον χρόνο. Γκρός, σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να το ευχηθώ καλή τύχη, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Έτσι και και ο καλύτερος Βέλγος εδώ πέρα θα, θα, απελπιστεί προσπαθώντας να βρει ένα συμβιβασμό. Αλλά ένα θα ήθελα να πω, όταν μιλάμε για ασφάλεια νομίζω πως υπάρχει ε, συνένεση δεύτερον για τις αεροδυναμικές βελτιώσεις και εδώ πέρα νομίζω πως μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε και όταν μιλάμε για τη μετατόπιση θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Όποιος θέλει να πάει από το α στο β και δεν υπάρχει σιδηρόδρομος, τίθε το ερώτημα πώς μπορούμε να το οργανώσουμε καλύτερο. Να φτιάξουμε σιδηρόδρομο ή να μετατοπίσουμε το εργοστάσιο. Δηλαδή, μην το ξεχνάμε. Εντάξει, υπάρχει μετατόπιση όπου υπάρχει η δυνατότητα. Αλλά γιατί δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή η μετατόπιση στο σιδηρόδρομο παρά το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση βλέπουμε πως δεν συμβαίνει αυτό το οποίο ελπίζουμε γιατί υπάρχει και θέμα υπηρεσιών και πολλών άλλων πραγμάτων. Οπότε έχει δίκιο εδώ πέρα η κυρία Κορίν Βόρτμαν Κόλ. Δηλαδή ε, απαγορεύεται στις ε, πόλεις ε, ουσιαστικά να γίνει κάτι τέτοιο. Έχετε Επίσης για μένα είναι ακατανόητη η συζήτηση για τις διασυνοριακές μεταφορές. Οπότε, τι θα γίνει, θα υπάρξει ένα δίκτυο περιορισμένο στην Ευρώπη εκτός ε, αστικών κέντρων. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συνένεση πρώτα μεταξύ μας και μετά με τις ε, υπόλοιπες ομάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι τηρήσατε και το χρόνο. Λοιπόν, ο κύριος Καραμίτσος τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας διαφωτίσει, θα μας πει τις πρώτες του σκέψεις. Κύριε Καραμίτσο. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιστρέψτε μου να χρησιμοποιήσω κάτι που είπε ο κύριος Μπαχ. Είπε ότι ζούμε στον 21ο αιώνα. Και βλέπω εδώ τις συζητήσεις ε, του 20ου αιώνα, 30 χρόνια πίσω, να επαναλαμβάνονται τώρα στον 21ο αιώνα. Χρησιμοποιείται αυτός ο όρος ε, τερατώδη οχήματα. Τώρα χρησιμοποιούμε το gigaliners και τα μέγα οχήματα. Παρακαλώ, η πρότασή μας δεν αφορά ούτε γίγαντες, ούτε τέρατα, ούτε τέτοια πράγματα. Η πρότασή μου είναι πώς θα πρασινίσουμε και θα κάνουμε πιο ασφαλή τα οχήματα, όπως είπαμε και τον Απρίλιο, όταν ξαναπήραμε το λόγο ενώπιον της Επιτροπής σας. Και το κύριο θέμα μας δεν είναι οι διασυνοριακές ε, ε, η διασυνοριακή κυκλοφορία. Η όλη συζήτηση τη διασκέδασα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι να εξαίρω τα πάθη μεταξύ των κρατών μελών. Πράγμα που είχε συμβεί και πριν από από 30 χρόνια όταν υιοθετήθηκε η πρώτη οδηγία. Δυστυχώς τότε είχα και μαύρα μαλλιά και ήμουν και νέο και ωραίο. Τέλο πάντων. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον κύριο Λάγκφιλντ. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Έχετε συμπεριλάβει πολλές θετικές εξελίξεις. Έχετε και κάποιες ε, τροπολογίες που συνιστούν βελτιώσεις και θα τις στηρίξουμε. Για παράδειγμα, η τεχνολογική ουδετερότητα, με την αύξηση του βάρους, ε, τα εναλλακτικά καύσιμα. Πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Η συμπερίληψη των αεροδυναμικών ε, δοκιμών, η τροπολογία 32. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που αμφισβητούν τον στόχο της αναθεώρησης και τις οποίες η τροπολογία νομίζω δεν μπορεί, η Κομισιό νομίζω δεν μπορεί ε, να υποστηρίξει. Ε, για παράδειγμα η 20, τροπολογία 20, γιατί τα 50 εκατοστά ήδη περιλαμβάνονται στη διαδικασία εγκρίσεων. Αλλά η όλη έρευνα που έχει γίνει από τον κλάδο έχει δείξει ότι τα πρόσθετα ωφέλη μπορούν ε, ε, να, μπορούμε να έχουμε αν πάμε και παραπάνω. Ε, με τα πτερή για αυτά που υπάρχουν πίσω. Δεν συμφωνώ ότι μπορούμε να πάμε στις συνδυασμένες μεταφορές. Ε, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν υλικά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί πράγματι με, με το μπροστινό και το πίσω μέρος των φορτηγών με τις τροποποιήσεις που έχουμε επιφέρει, έχουμε μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με υψηλά περιβαλλοντικά ωφέλη και καλύτερη ασφάλεια. Γιατί και οι συνθήκες ζωής για τον οδηγό και για τους ε, πεζούς ε, βελτιώνονται με τον ε, σχεδιασμό του προστινού μέρους των οχημάτων. Βελτιώνεται η αεροδυναμική, βελτιώνεται η κατανάλωση ενέργειας και κατ' επέκταση βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδεση. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία της έκθεσής μας όχι διασυνοριακή κυκλοφορία. Εάν τα κράτη-μέλη συμφωνούν πάνω στο θέμα αυτό, ας το κάνουμε αύριο, ας υιοθετήσουμε ένα νομοθέτημα και αύριο κιόλας. Ε, δεν ξέρω με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο τι συμβαίνει με τα ψηλότερα οχήματα σε τεστ που έχουν γίνει, σε δοκιμές που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, στις κάτω χώρες, στη Γερμανία. Ε, οι έρευνες που έχουν γίνει πιστοποιούν τα, τις βελτιώσεις και δεν, και δεν μιλούμε για την αύξηση βάρους, έτσι. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και την αύξηση βάρους, αλλά εμείς συζητούμε μόνο το θέμα της αλλαγής των διαστάσεων. Είναι ένα παράδειγμα νομοθετήματος Νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα με τις υποχρεωτικές διατάξεις περί ασφαλείας. Είμαστε υπέρ. Αλλά, αλλά τα θέματα αυτά συζητώνται σε άλλα επίπεδα. Εμείς ξεκινούμε με την ιδέα να συμπεριληφθούν σε εθελοντική βάση όλες αυτές οι συσκευές βελτίωσης της ασφάλειας, αλλά για να γίνουν ε, υποχρεωτικά πρέπει να συνεννοηθούμε και με άλλους, με άλλες πλευρές. I Unfortunately, Δυστυχώς το, το όλο ζήτημα διασυνοριακής κυκλοφορίας ε, οφείλεται σε παρανόηση νομίζω. Δεν μιλούμε εδώ, δεν γίνεται λόγος εδώ ε, για διασυνοριακή κυκλοφορία μεγάλων, πολύ μεγάλων φορτηγών και δυστυχώς πολλές τροπολογίες με αυτό ασχολούνται. Δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά των φορτηγών μεγαλύτερων διαστάσεων, μεγαλύτερου μήκους. Απλώς συμπεραίνουμε ότι τίποτε στην τωρινή μας οδηγία δεν υπάρχει που να εμποδίζει τα φορτηγά αυτά να κινούνται μεταξύ ε, των κρατών μελών εφόσον τα κράτη-μέλη εγκρίνουν την κυκλοφορία τους. Τώρα, τα θέματα αυτά βέβαια πρέπει να τύχουν και τη έγκριση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, να μην το ξεχνούμε αυτό. Ε, θα ήταν παράλογο να πούμε ότι ένα όχημα το οποίο την χάνει της έγκρισης δύο ή τριών κρατών μελών δεν μπορεί να διασχίζει τα σύνορα. Ε, νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι μια τέτοια προσέγγιση στους λαούς μας και στα κράτη και νομίζω ότι σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας πρέπει να, να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι σκέφτονται οι πραγματικοί πολίτες μας που οδηγούν στο δρόμο. Φοβάμαι ότι παρακολούθησα όλη τη συζήτηση για τα βαρέα και μακρά οχήματα Εφόσον όμως αυτό δεν ήταν το θέμα των συζητήσεων στην Κομισιόν, να σας πω και τα εξής, κύριε Πρόεδρε. Όλες οι δοκιμές που έχουν γίνει στην Αλλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, έχουν δείξει, έχουν αποδείξει ότι τα οχήματα αυτά έχουν ε, μόνο ωφέλη να φέρουν, όχι αρνητικές συνέπειες. Οπότε παρακαλώ να συζητήσουμε και να δούμε την έκθεση, για να, έτσι ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα πράγματα αυτά στις τελικές συζητήσεις. Και κάτι άλλο. Κοιτάξτε ξανά παρακαλώ τη γνωμοδότηση της ε, ΕΚΟΣΟΚ, η οποία μάλιστα εγκρίθηκε και ομόφωνα και η οποία συμφωνεί με την πρότασή μας και θεωρεί ότι είναι η καλύτερη συμβιβαστική λύση σε περίοδο κρίσης όπου θέλουμε να βελτιώσουμε και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας μην ξεχνούμε ότι τα φορτηγά αυτά ε, χρησιμοποιούνται και στις εξαγωγές για τη βιομηχανία μας και πρέπει να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να, να αναπτύσσουν το σχεδίασή τους, να επιφέρουν τεχνολογικές καινοτομίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Καραμίτσο. Πράγματι ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας. Σε αντίθεση με πάρα πολλούς ε, σε αυτή την αίθουσα πράγματι δεν έχετε ε, έτσι πάρα πολύ ε, ιδέες επηρεασμένε ε, από κάποιες ε, προκαταλήψεις. Βλέπω όμω ότι κάποιο θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ναι, μια σύντομη ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Από την αξιολόγηση των μεγάλων αυτών φορτηγών υπάρχουν αποτελέσματα για την ειδική κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο και χιλιόμετρο σε σχέση με τα κανονικά φορτηγά και από την τεχνολογική πλευρά της ανάπτυξης αυτών των ε, μεγάλων φορτηγών των Gigaliners όσον αφορά τις τρεις πτυχές, δηλαδή βελτίωση της σχέσης μάζας ε, προς απόδοση, τον συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης και την ε, αντίσταση κύλησης. Όταν μιλάμε δηλαδή για, για βελτίωση υπάρχει όντω. Γιατί δεν έχει νόημα να λέμε τα κάνουμε όλα μεγαλύτερα, μακρύτερα κτλ. Ε, δεν έχει αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα κατανάλωση ανατόνο και χιλιόμετρο. Αυτό με ενδιαφέρει σε σύγκριση με τα κανονικά φορτηγά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ε, κάπως μεσαία ερώτηση. Σύντομη απάντηση παρακαλώ. Νομίζω υπάρχουν πληροφορίες, έχουμε κάνει αξιολόγηση αντικτύπου ε, προτείνω να έρθουμε σε άμεση επαφή, να σας δώσω τα λεπτομερή νούμερα και, και στον εισηγητή νομίζω. Γιατί ε, νομίζω πως πρέπει να συνεχίσει η συζήτηση με τον εισηγητή σε πνεύμα θετικό. Σας ευχαριστώ. Πριν τελειώσουμε θα ήθελα να δώσω στον εισηγητή την ευκαιρία να πει κάποια πραγματάκια ακόμα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πάρα πολλά. Αλλά Λέτε πως πρέπει να προσέχει το Ευρωπαϊκό... Ακούστηκε πως πρέπει να προσέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που τελευταία έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις η Κομισιόν. Ε, σκέφτεται δηλαδή το να απαγορεύσει το ασφράγιστο ελαιόλαδο και το σανέλ νούμερο 5 κτλ. Να μην οδηγηθούμε σε κάτι ανάλογο και σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βόρτμαν Κόλ και τους συναδέλφους από το Λουξεμβούργο που με βοήθησαν πάρα πολύ εδώ πέρα. Εγώ θα ε, ήθελα πράγματι να έχει υπάρξει καλύτερη προετοιμασία. Θα ήθελα αναλυτικότερη μελέτη αντικτύπου. Γιατί έτσι θα είχαμε ε, επιστημονικά δεδομένα όχι μόνο από τον κάθε λομπίστα, έτσι, γιατί υπάρχει μια εμπειρογνωμοσύνη του ενός και μετά μια από την άλλη πλευρά. Και είτε όλοι έχουν δίκιο είτε δεν έχει κανένας. Αν είχαμε λοιπόν κάτι έγκυρο θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε το να κάνουμε ή να μην κάνουμε το χ ή το ψ πράγμα. Τώρα δεν γίνεται, τέλος πάντων με αυτά που έχουμε θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα. Να πω τώρα κάτι αν μου επιτρέπετε, αναφέρθηκε η αρχή της επικουρικότητας από κάποιους ε, συναδέλφους. Γιατί λέτε πώς μπορούν να ξεπεραστούν κάποια εθνικά μέγιστα όρια. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν ανώτατα όρια τα, ε, τα οποία θα ξεπεραστούν, γιατί να μην συμβαίνει και το αντίστροφο. Να πει μια χώρα εγώ θέλω μόνο 38 τόνους. Έτσι πρέπει να υπάρχει και κάποια δικαιοσύνη εδώ πέρα, να, υπάρχει να ισχύουν τα ίδια για όλους και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ε, εάν ξεπερνιούνται σε κάποιες χώρες ε, το ζήτημα είναι το τι γίνεται όντως και αν ε, το αναγνωρίζουμε de facto. Γνωρίζω ήδη πως ε, εάν περάσει η έκθεσή μου όπως έχει θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Πρέπει πράγματι να το συζητήσουμε, δεν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα όπου θα πρέπει να περιορίσει τη διασυνοριακή κίνηση η Μεγάλη Βρετανία με την Ιρλανδία, έτσι. Εδώ πέρα συμφωνώ με τους συναδέλφους. Τέλος, για να μην σας φάω και πολύ χρόνο, να σας ευχαριστήσω για την καλή συζήτηση, τις επικοδομητικές ε, προτάσεις. Νομίζω πως ε, θα καταλήξουμε τελικά σε κάτι λογικό. Mm, να πω στον Πίτερ Φαντάλ, ναι, όλοι θέλουν βελτίωση, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Έτσι. Νομίζω πως ε, εδώ πέρα μπορούμε να, συμφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους όσους ε, συμμετείχαν στη συζήτηση. Προθεσμία για τροπολογίες είναι στις 5 Δεκεμβρίου Εμείς ε, δίνουμε δώρα στις 5 Δεκεμβρίου στην Ολλανδία. Τα δώρα αυτά θα είναι τροπολογίες σε αυτή την περίπτωση. 5 Δεκεμβρίου λοιπόν, 12 η ώρα. Αυτά για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. akkoord. Σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω στην ημερήσια διάταξη. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Στην αίθουσα. Συνεχίζουμε με το σύστημα e-call στα ΙΧ. Ο κύριος Ντεμπάκερ είναι ο εισηγητής ο οποίος έχει τον λόγο. Θα ξεκινήσει αυτός λοιπόν και μετά θα ακολουθήσουν οι σκιώδες εισηγητές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δύο θέματα σε ένα. Το ένα αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή ενός διαλειτουργικού συστήματος e σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη έχουμε και γνωμοδότηση ε, προς την Επιτροπή Εσωτερικής ε, Αγοράς ε, για την έγκριση τύπου για τα συστήματα τα ενσωματωμένα και θα τα δούμε αυτά μαζί η, έκθεσή μου, η θέση μου να την ξεκαθαρίσω. Συμφωνώ 100% με την πρόταση της Κομισιόν για το να είναι υποχρεωτικό το σύστημα από 1η Οκτωβρίου 2015 για όλα τα καινούργια οχήματα. Σήμερα 1% των οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα e-call. Είναι κάτι το τελείως ε, εθελοντικό και η εθελοντική προσέγγιση οπότε φαίνεται δεν λειτουργήσε. Η αυτόματη κλίση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο γρήγορη επέμβαση των υπηρεσιών πρώτης ε, βοήθειας. Οπότε πρέπει να επικρατήσει ασφάλεια σε, σε περίπτωση ατυχήματος κάθε λεπτό μετράει και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να διηγηθούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ελπίζω λοιπόν να μην έχουμε πάλι άλλες ε, καθυστερήσεις. Τι προτείνουμε λοιπόν Πρώτον βεβαίως υπάρχει ήδη η υπηρεσία 112, θα πρέπει να υπάρχει και η σωστή λειτουργία των ε, σημείων ε, των υπηρεσιών ασφαλείας. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια επένδυση, αλλά οι επενδύσεις αυτές νομίζω θα είναι ελάχιστες. Θα πρέπει επίσης να ε, απλοποιηθεί και ίσως να αναβαθμιστεί η σχετική υποδομή. Εδώ πέρα ζητάω, όπως και η Κομισιόν, ε, η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη να κάνουν μια εξαρτία ενημέρωσης για το νέο σύστημα και τις δυνατότητές του. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα να υπάρξει ένα φιλτράρισμα στις κλήσεις ε, τις αυτόματες και τις μη αυτόματες κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Επίσης ε, το να είναι αξιόπιστος ο εντοπισμός του σημείου του ατυχήματος είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. και βεβαίω είναι σημαντικό για όλες τις κλήσεις ε, ανάγκης. Για το δεύτερο θέμα τώρα, για την έγκριση τύπου, συμφωνώ με το πεδίο εφαρμογή που προτείνει η Κομισιόν. Η Κομισιόν μπορεί να διερευνήσει το εάν θα πρέπει να επεκταθεί και στα δίκυκλα, τα βαρέα φορτηγά και τα λεωφορεία. Επίσης, ε, η έκκληση που απευθύνεται στους κατασκευαστές ε, να υπάρξει ενσωμάτωση των υφιστάμενων συστημάτων στο σύστημα το προτινόμενο. Μια ανοιχτή πλατφόρμα νομίζω είναι το καλύτερο σύστημα, αλλά νομίζω πως απαιτείται, ε, μια, απαιτείται περισσότερη έρευνα. Και νομίζω μπορούμε να αφήσουμε την πρόταση Κομισιόν ως έχει για να εφαρμοστεί γρήγορα και να ενσωματωθεί το σύστημα σε όλα τα νέα οχήματα. Επίσης σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον ορισμό της ηλεκτρονικής κλίσης και βεβαίως ε, υπάρχει και συζήτηση με τους διαφόρους κατασκευαστές που προσφέρουν ήδη τα δικά τους τέτοια συστήματα και δεν σκοπεύουμε να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι προσφέρουν ήδη μια τέτοια υπηρεσία. Έτσι, είναι μια προσθέμενη αξία για πολλούς οδηγούς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στους οδηγούς, στους καταναλωτές να μπορούν να διαλέξουν και να ε, ξεκαθαρίζουμε πως ε, υπάρχει ως βασικό σύστημα από 1η Οκτωβρίου 2015 το σύστημα κλήσης του 112 το οποίο θα προσφέρεται σε όλους. Οπότε ε, να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά μεταξύ των ε, διαφορετικών συστημάτων και βεβαίως να υπάρχει και τεχνολογική ουδετερότητα όσον αφορά τα υφιστάμενα τέτοια συστήματα. Και εδώ πέρα συμφωνήσαμε τους κοιόδης ηγητές, πρέπει να δούμε με τον κλάδο πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λογική πρόταση. Τέλος, προστασία της ιδιωτικής ζωής, πάρα πολύ σημαντικό, να μην υπάρχει κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει το σύστημα αυτό να είναι ενυπνώση και Επίσης, στην περίπτωση στην οποία επιλεγεί ένας ε, τρίτος ε, κατασκευαστής, να υπάρχει σαφής ενημέρωση του καταναλωτή. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα σημεία της εκθεσής μου, αλλά αναμένω και την ε, συζήτηση που θα έχουμε με τους σκιοδησηγητές και τους συναδέλφους για να μπορέσουμε 1 Οκτωβρίου 2015 να έχουμε πράγματι εισαγωγή αυτού του συστήματος. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά για την παρουσίασή σας. Περνάμε τώρα στους και ηγητές. Και ο Σκόχ έχει το λόγο. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι σημαντικό ε, να ξέρουμε πόσο χρόνος πιέζει. Κάθε μήνα που χάνουμε, κάθε μήνα που καθυστερούμε, σημαίνει πως χάνονται οι ανθρώπινες ζωές. Έτσι, μέχρι, πολλοί λένε μέχρι και 100 ζωές. Υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα σε πολλές ε, εταιρείε. Ε, δεν είναι σύστημα άνεσης ή βοήθειας ε, του οδηγού. Είναι σύστημα το οποίο ειδοποιεί αμέσως τις υπηρεσίες βοήθειας για να έρθει ως το δυνατόν πιο, πιο γρήγορα επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Απαιτείται λοιπόν, απαιτούνται λοιπόν κάποια ελάχιστα δεδομένα κάτι το οποίο χρειάζονται βεβαίως και οι τρίτες ε, εταιρείες και οι τρίτοι κατασκευαστές. Περαιτέρω δεδομένα όμως από τα απολύτω απαραίτητα, απαραίτητα δεν πρέπει να είναι διαθέσιμα. Έχουμε λοιπόν ε, ως τρίτους ε, και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων αλλά και τις λέσχες οδικής βοήθειας κτλ. Βεβαίως εδώ πέρα θα πρέπει για τα παραπάνω δεδομένα, πέρα από τα πολύ απαραίτητα, να υπάρχει έγκριση του οδηγού και μην ξεχνάμε ότι από ένα σημείο και μετά είναι δικά του ιδιωτικά και δεύτερον πρέπει να υπάρχει βεβαίως και μία κάποια προστασία και βεβαίω να υπάρχει ένα δικαίωμα, να έχουν περιορισμένοι άνθρωποι ένα δικαίωμα πρόσβασης. Ε, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί, Ποιο μπορεί να δει αυτά τα δεδομένα. Επίσης μην ξεχνάμε πως οι κλήσεις ανάγκης ε, είναι παντού δωρεάν, ε, δεν κοστίζουν και έτσι πρέπει να είναι ενώ τα ιδιωτικά συστήματα βοηθείας ε, έχουν τη δυνατότητα και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιπλέον να προσφέρουν κάποιες άλλες υπηρεσίες. Αλλά αυτό πάντα με βάση μία σύμβαση μεταξύ του πολιτή και του αγοραστή ή του χρήστη του οχήματος. Τώρα δεν ξέρω, πώς δεν ξέρω δεν είμαι σίγουρος για το αν θα πρέπει να υπάρξει υποχρέωση επανεξοπλισμού των παλαιότερων οχημάτων. Βεβαίω δεν θα εμποδίσουμε και κανέναν να αναπτύξει άλλες έξτρα συσκευές ε, οι οποίες θα λειτουργούν. Νομίζω πρέπει να τις δεχτούμε και να μην τις απαγορεύσουμε σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πρέπει να καταλήξουμε σύντομα σε ένα δεσμευτικό αποτέλεσμα για να υπάρξει επιτέλους η ηλεκτρονική αυτή κλίση. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές, κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα γνωρίζετε όλοι ότι πρόκειται για μια μακρά διαδικασία για την εναρμόνιση του διαλειτουργικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το e Είναι στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2005. Δεν είναι από τις πρώτες προτεραιότητες, αλλά είναι σημαντικότατο ζήτημα. Χρειάζεται λοιπόν κατά προτεραιότητα δράση για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη ενός συστήματος e στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική που βασίζεται σε μια κατεξοχήν ρυθμιστική προσέγγιση προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις του τηλεπικοινωνιακού συστήματος και του EPS ε, των ε, σημείων ε, το e-call συνδυάζεται με τους νέους στόχους που έχουν ε, εισαχθεί στο σύστημα για την οδική ασφάλεια και τις προτεραιότητές του με συγκεκριμένους στόχους για το 2011 που υπολογίζει ότι υπάρχουν 1,1 εκατομμύρια οδικά ατυχήματα στους δρόμους της Ευρώπης ετησίως. Επίσης, ε, υπάρχει οικονομικό βάρος για τους φορείς με 2,4 δις ευρώ ετησίως Βεβαίως κάθε ανθρώπινη ζωή μετράει. Οι πολίτες θα μπορούσαν να είναι προστατευμένοι και 4.000 ζωές να ε, σώζονται ε, συνέχως ε, με την χρήση του συστήματος Κατά πρώτον, λοιπόν, να εκφράζω την εκτίμησή μου προς τον εισηγητή για την έκθεση του. Ήταν πολύ σημαντική η επικοινωνία που είχαμε στις επανειλημμένες συναντήσεις μας αλλά ως προς την ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος η κόλλη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναθ, ε, αναγνωρίζω για το 7α ε, το 7-8 μάλλον τη σημασία της ε, ευαισθητοποίησης του κοινού. Επίσης, όπως είπε η συνάδελφος Όλγα στην γνωμοδοτησή της, το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί διαφορετικοί πολίτες, να, ε, οι διάφοροι μαλλοπολίτες ανακατηγορία να καταβάλουν αντίτιμο. Το πλέον περίπλοκο ζήτημα βεβαίως έχει να κάνει με τις απαιτήσει αντιδότησης για την ανάπτυξη του συστήματος e Συμφωνώ πολίτες με τον εισηγητή, την Όλγα, και την τροπολογία της 3 των ιδεολογική σκέψη 7, ότι θα πρέπει το e να συνδυαστεί με άλλες ρυθμιστικές προσεγγίσεις που έχουμε, γι' αυτό τα συζητάμε και στις συναντήσεις των σχεδόν συγκητών, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω να με ακούτε, να προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα και μελέτη αντικτύπου. Επίσης θα πρέπει να γίνουν αυτά παράλληλα, γιατί το 18 συγκεκριμένα, το 2018 είναι υπερβολική φιλοδοξία. Στο 7 για την αιτιολογική σκέψη 9 το e-call θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε διατηρητική βάση και ε, ανοιχτή στην πρόσβαση πλατφόρμα, αλλά τυποποιημένη. Φαντάζομαι σε αυτό θα συμφωνείτε. Επίσης, η στρατηγική προσέγγιση είναι πολύ καλή από την πλευρά του σύγκριτη. Και θα συμφωνήσω με την Όλγα στι τροπολογίες 14 και 20. Αντί να διατηρήσουμε τα ε, άρθρα 3,2 της Επιτροπής, τα αρχικά άρθρα, θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα εντός των οχημάτων ε, και να το ορίσουμε με σαφήνεια. Επίσης πρέπει να έχουμε σημαντικ... Ε, βασικούς στόχους για την παρακολούθηση του πώς λειτουργεί το συστημα ECOL. είναι ένα δημόσιο σύστημα πανευρωπαϊκό το οποίο θα βασίζεται στο 112 θα πρέπει να λειτουργεί σε όλα τα ευρωπαϊκά οχήματα από την 1η Οκτωβρίου 2015. Τα κάτι μελη θα πρέπει να οργανώσουν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού το αργότερο στην 1η Οκτωβρίου 2015 και πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στην ε, πανευρωπαϊκή κλίμακα και τη λειτουργικότητα του e βάσει των προδιαγραφών που εμείς οι ίδιοι έχουμε ε, ε, ορίσει. Δεν, θα ήταν, ε, δεν είναι περίεργο αυτό. ω προς την προστασία των καταναλωτών όλων των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στο σύστημα e παντού, οπότε γεωγραφικώ θα πρέπει να καλύπτεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, όλοι οι ε, αυτοκινητοπαραγωγοί θα πρέπει να κατανοήσουν και θα πρέπει να τους υποχρεώσουμε με ρυθμίσεις ότι όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν θα πρέπει να έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές για να αναγνωρίζουν το σύστημα οίκων και να το χρησιμοποιούν. Θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει ο τεχνικός εξοπλισμός εντός του οχήματος και να έχει καλυφθεί από την τελική τιμή του οχήματο. Η ασφάλεια δεν θα πρέπει να παίζεται στα έξτρα στοιχεία θα πρέπει να είναι η τιμή προσιτή για τους Ευρωπαίους οδηγούς. Ευχαριστώ πολύ για την εξωτερική μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ και εγώ. και για την ε, παρέμβασή σας ε, και για την ε, στήριξή σας. Δεν βλέπω τους υπόλοιπους οικειώδες ηγητές, οπότε θα δώσω λόγο στην κυρία Σενάλοβα. Děkuji, eh, pane předsedající. Já dnes eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να να πω ότι σήμερα θα παρουσιάσω στην Επιτροπή IMCO την δική μου, το δικό μου σχέδιο έκθεση για, για το σύστημα ECOL. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω ότι είναι πολύ καλή η συνεργασία μα με την ΟΠΤΕΠΗ, ΤΡΑΝ και τον ΕΣΥΤΗ σα. Βλέπουμε εδώ το σχέδιο έκθεσης να οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να ακολουθεί τη θέση που υποστηρίξα και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Θα αναφέρω ορισμένες μόνο τροπολογίες ε, για τις οποίες έκανε επενιγμούς ο κ. Ντεμπάκερ. Ένα πράγμα με το οποίο θα συμφωνήσω είναι οπωσδήποτε η τροπολογία 2 που αφορά τις ε, εκστατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωση για το σύστημα Όντως, θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν το γεγονός ότι τέτοια συστήματα διατίθενται και ότι έχουν προστιθεμένη αξία για την ζωή τους και την ασφαλεία τους. Δεν τα γνωρίζουν επαρκώς αυτά οι πολίτες. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξουν εξτατείες ευαισθητοποίησης. Θα ήμουν όμως ε, περισσότερο διστακτική με την τροπολογία 3 το να εντοπιστεί ένα όχημα που χρησιμοποιεί κινητά, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι κάτι εφικτό μεν, αλλά θα πρέπει εδώ να επικεντρωθούμε περισσότερο στο να εισάγουμε ένα σύστημα e-call ανεξαρτήτως από τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Όχι να προσθέσουμε και άλλες πτυχέ που να ε, ε, επιφέρουν επιπλοκές στην ε, όλη κατάσταση του συστήματος. Θα καθυστερήσουμε έτσι. Σε ό,τι αφορά την προτάση γνωμοδότηση θα συμφωνήσω με τις περισσότερες από τις προτινόμενες παρατηρήσει του κειμένου, αλλά να πω ότι υποστηρίζω την τροπολογία 2, δηλαδή ότι από το 2015 να είναι εξοπλισμένα με το σύστημα e τα περισσότερα οχήματα, όσο δυνατόν περισσότερα, και να υπάρχουν και συστηματικοί τεχνικοί έλεγχοι όπως αναφέρεται στι τροπολογίε 5 και 13. Είναι κέρια σημασία. Παρομοίω με τις εκθέσεις αξιολόγηση που θα πρέπει να συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευρύνοντα κάπως το πεδίο του κανονισμού όπως αναφέρει και η τροπολογία 16. Το θέμα είναι εάν αυτά θα ξεκινήσουν το 2016 ή το 2018 αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχω καμία αντίρρηση ως προς το σχέδιο έκθεσης και πραγματικά ανυπομονώ να προχωρήσει με βήμα ταχύ η έκθεση αυτή, να εγκριθεί γρήγορα και μάλιστα εντός της θητείας μας, ώστε το σύστημα e-call να μπορέσει επιτέλους να λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου 2015. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πάλι τον κύριο Καράμου ακούσουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που αυτό το θέμα δεν προκαλεί τόση διχογνωμία όπως το προηγούμενο. Ε, φαίνεται ότι όλα τα κράτη-μέλη κατανοούν πως πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως οι προτάσεις μας βασίζονται ε, στην ε, έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, του κύριου Κόχ και άλλων, στην έκθεσή σας καλέσατε την ε, Κομισιό να υποβάλει μια πρόταση για να εξασφαλιστεί η υποχρεωτική επέκταση του συστήματος υποχρεωτικής κλήσης μέσω του αριθμού 112 σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να αναβαθμίσουν τους μηχανισμούς ανταπόκρισης της κλήσης έκτακτης ανάγκης, βελτιώνοντας τις ε, ε, εθνικές υποδομές και ανοίγοντας την πρόσβαση σε όλους. Αυτό είναι το νόημα των προτάσεων ε, που υπέβαλε η Κομισιόν. Τα αυτοκίνητα λοιπόν θα καλούν υποχρεωτικά αυτόν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σύγκρουσης. Επιτρέψτε μου να πω εν συντομία, και μερικοί το αναφέρατε κιόλα, ότι κάθε λεπτό μετά από ένα ατύχημα, γιατί το 50% ε, των θανάτων επέρχονται λεπτά μετά από το ατύχημα. Ε, με όλες τις μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να μειωθεί κατά 40% σε αστικές περιοχές και μέχρι και 50% στην Ήπεθρο και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ήπεθρο γιατί το 60% των θανάτων ε, συμβαίνουν γιατί χρειάζεται κατά μέσο όρο 10 λεπτά για να προσέλθουν ε, οι υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας. Κατανοούμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει το e Αυτή τη στιγμή δυστυχώς η δίσδυση είναι πολύ χαμηλή. Οι ιδιώτες πρέπει να το κάνουν, οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι εκείνες που πρέπει να το συμπεριλάβουν στα αυτοκίνητα. Μετά από προσπάθειες 10 ετών, δυστυχώς μόνο το 0,7% των οχημάτων είναι φοδιασμένα με ένα σύστημα αυτόματης κλήσης, e-call παρά τα ωφέλη των άλλων συστημάτων που υπάρχουν, των συστημάτων ανταπόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ε, η κάλυψη είναι πολύ μικρή και Όπως είπαμε λοιπόν, μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 θέλουμε όλα τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με τέτοιο, τέτοιους μηχανισμούς. Είναι μια λύση εύκολη, φτηνή. Το κόστος αυτών των συσκευών είναι περίπου 14 ευρώ νομίζω για όλους και είναι ο μόνος τρόπος εξασφάλισης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών τέτοιων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας όλη τον κύκλο ζωής των οχημάτων. Ε, και βεβαίω θα υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο ανταπόκριση, ε, πλήρω τυποποιημένο που θα λειτουργεί εύρυθμα. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν εκείνα με τον τρόπο που νομίζουν καλύτερο το σύστημα ανταπόκριση. Μπορούν να έχουν ένα σύστημα φιλτραρίσματος των κλήσεων για έτσι να αποκλείονται οι κλήσεις που δεν είναι πραγματικά έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει τώρα το θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε εξασφαλίσει με την πρότασή μας ότι το σύστημα e-call θα σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα προστατεύει την προσωπικότητα των πολιτών και ελπίζω ότι αυτό θα περάσει και στο τελικό κείμενο. Για τις ε, τροπολογίες τώρα που έχουν προταθεί, νομίζω ότι μπορούμε να, να τις δεχτούμε τις περισσότερες. Ε, θα ήθελα λίγο να αναδείξω κάποιες πτυχές που δεν είναι τόσο σαφείς. Έχουμε τον Γαλιλαίο. Μία από τις προτεραιότητες μας στο σύστημα Γαλιλαίος είναι να χρησιμοποιείται στο μέλλον για πολλές εφαρμογές και μία από αυτές τις εφαρμογές είναι στις μεταφορές. Σύστημα που να, συστήματα που να βελτιώνουν την ε, αποτελεσματικότητα, το περιβάλλον και την ασφάλεια στις μεταφορές. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την διάσταση και πάνω σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Ντεμπάκερ και την τροπολογία και υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρχει αυτή η ιδέα, το GNSS που θα περάσει στο Γαλιλαίο στο μέλλον. Παρόλο που είναι δύσκολο να το εισάγουμε μέχρι το 2015, αλλά θα πρέπει τα συστήματά μας να είναι ανοιχτά έτσι ώστε να το ενσωματώσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, έτσι ώστε η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα να εξασφαλιστούν. Και στις υπηρεσίες Γαλιλαίος υπάρχουν διατάξεις που θα μας το επιτρέψουν αυτό. Μην το χάνουμε αυτό από τα μάτια μας. Και το λέω αυτό και προς τους συναδέλφους μου στη Γενική Διεύθυνση ε, Enterprise. Να χρησιμοποιήσουν αυτό που υπάρχει και να διατηρήσουμε το πνεύμα μας ανοιχτό. Ε, λίγο πολύ αυτό ήθελα να τονίσω και να πω και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον εισηγήτη για να βελτιώσουμε το κείμενο όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σα και την αντίδραση. Κύριε Ντεμπάκερ, θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Σύντομα. ορίζω τα θετικά σχόλια των συναδέλφων σχόλια που έχουν γίνει και σε άλλε περιστάσει. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε καλέ συμβαστικέ λύσει, να βελτιώσουμε το κείμενο, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε σύντομοι και γρήγοροι. Να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου 2015. Νομίζω οι πολίτε μα αξίζουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη θετική τους στάση, τα επικοδομητικά του σχόλια και ανυπομονώ για τη μελλοντική μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Θα πάμε γρήγορα. Πρόταση, προθεσμία για τροπολογίες 13 ε, Νοεμβρίου το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα. πρέπει να είναι εδώ ο κύριος Ρούτε. Πέντε λεπτά. Ωραία. Ένα διάλειμμα πέντε λεπτών. Συνεχίζεται η συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που ήρθε ο κύριος Ρούτε για να μας μιλήσει για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Θα λάβετε λοιπόν πρόταση στον λόγο και μετά οι συγητές από την Επιτροπή μας. Ο κύριος Μαρινέσκου ήρθε ήδη και μετά βεβαίως οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Ρούτε. Έχετε τον λόγο. Thank you very much, uh, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας. Προσπαθώ να έρχομαι από καιρού εις καιρών και είναι μεγάλη χαρά μου που σας παρουσιάσω την πρόταση ε, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό 2 συν. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό για μένα είναι να ακούσω τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, και να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Δεν ήταν εύκολη επιλογή για τον Αντιπρόεδρο Κάλλας να υποβάλει αυτή την πρόταση. Και ονομάζεται ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 2 συν, ε, γιατί αποτελεί συνέχεια ε, της πρότασης για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό που συζητήσαμε πριν από μια διετία περίπου. Επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε την προσέγγιση μας, την οποία έχουμε αναπτύξει, για, να, για την αντιμετώπιση των ε, φυσικών μονοπωλίων μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Πέρυσι στην ε, Λέμεσό έγινε ένα συνέδριο και είχατε αρκετοί από εσάς ήσασταν εκεί. και και από την πλευρά της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ε, πολλές φωνές ακούστηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Τα πράγματα μάλλον δεν λειτουργούν καλά. Έτσι υπόθηκε τότε και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που ο Αντιπρόεδρος είπε εντάξει πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πριν να παρουσιάσω όλα τα επιχειρήματα για το γιατί δεν λειτουργούν τα πράγματα, ε, να πω ότι ε, εν μέρη σε συγκεκριμένους τομείς έχουν επιτευχθεί πρόοδοι και βελτιώσεις. Για πρώτη φορά σταματήσαμε την ετήσια αύξηση στο κόστος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας για πρώτη φορά. Επίσης, δημιουργήσαμε ένα ασφαλές ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο εν μέρη αποδίδει καρπούς και κινούμαστε ε, και στην υλοποίηση του τεχνολογικού πυλώνα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού μέσω, είτε, είτε μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών, είτε μέσω του manager, είτε μέσω των επεκτάσεων που συζητούμε. Αλλά νομίζω στην επιτροπή αυτή και και ένα μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου και αυτή η Επιτροπή συμφωνούν ότι η πρόοδος παρά είναι αργή και παρά είναι κερματισμένη. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός ο, ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Οργανισμός 2 ΣΥΝ στόχο έχει να, να κάνει τις ε, επισκευές στο προβληματικό, στον προβληματικό μηχανισμό και να, να σφίξει τις βίδες, αν θέλετε. Υπό αυτή την έννοια δεν πρόκειται για μια καινούρια πολιτική. Αυτό θα πρέπει να το πούμε σαφώς ευθύς εξ αρχής. Τι είναι λοιπόν αυτό που δεν λειτουργεί. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Στο προηγούμενο σχήμα ε, ε, Το προηγούμενο σχήμα ήταν πολλά υποσχόμενο, αλλά οι επιδόσεις του ήταν μόνο μερικώς επιτυχημένες. Για μόνο δεν επιτύχαμε την, ε, τον στόχο για την αποτελεσματικότητα του κόστους. υπάρχει η εξαίρεση για το ανεξέλεγκτο κόστος, η οποία οδήγησε σε μια κατάσταση όπου στην πραγματικότητα είχαμε πραγματικά κόστη τα οποία με το ζόρι συγκρατούμε. Επίσης δεν καταφέραμε να ορίσουμε τους στόχους ασφάλειας για τους οποίους συζητούσαμε το 2009. Δεύτερον, έχουμε τα λειτουργικά θέματα του εναέριου χώρου. Ε, τα λειτουργικά αυτά τμήματα αναπτύχθηκαν και θυμάμαι και τις διαπραγματεύσεις. Τα λειτουργικά αυτά τμήματα αναπτύχθηκαν ε, μέσα από συμφωνίες με τα κράτη-μέλη και επαφέθηκε στα κράτη-μέλη η ενοποίηση ε, του εναέριου χώρου. Ε, και τώρα τι έχουμε. Δίπλα σε αυτά τα blocks, τα λειτουργικά blocks, έχουμε νέα γραφειοκρατικά τέρατα τα οποία δημιουργήθηκαν. Έτσι, Διατηρούμε την, την παλιά εθνική προσέγγιση και δημιουργούμε ένα πρόσθετο στρώμα γραφειοκρατίας. Αυτό τελικά έγινε. Μερικές φορές αυτό οδήγησε τα κράτη-μέλη ε, σε μέτρα προστασίας του εισοδήματος των εθνικών τους παρόχων και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύονται και ε, τα μη αποτελεσματικά δρομολόγια. Τα κράτη-μέλη ισχυρίζονται ότι ο κανονισμός ε, είναι πολύ απαγορευτικός, ε, ότι περιλαμβάνει πολύ αυστηρές ρυθμίσεις. Εντάξει, μπορούμε να εισαγάγουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία στα λειτουργικά μπλοκ των εναέριων χώρων. θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε στον κλάδο τη δυνατότητα να αναδιοργανωθεί όπου αυτό είναι εφικτό. Και επιτρέψτε μου να, να είμαι πάρα πολύ σαφής. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, ε, βασικές υπηρεσίες, οι οποίες συνιστούν φυσικά μονοπόλια. Αλλά υπάρχουν και μη ουσιώδεις υπηρεσίες, όπου μπορούμε να είμαστε πιο καινοτόμοι, πιο αποτελεσματικοί, και μέσω των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων μπορούμε να επιτρέψουμε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων και των τελικών χρηστών. Και τέλος, ε, παραδόξως, η διαχείριση της αναέρειας κυκλοφορίας, και το ξέρετε ε, καλύτερα από μένα, αποτελεί έναν ξεχωριστό κόσμο και υπάρχει ελάχιστη πολιτική βούληση μεταξύ των κρατών μελών να παρέμβουν σε αυτόν τον κόσμο. Και το βλέπουμε αυτό όταν αναλύουμε τον αριθμό της ε, ρυθμιστικής εποπτείας που λαμβάνει η χώρα. Σε μεγάλο μέρος είναι αδύναμη και αναποτελεσματική η εποπτεία. Γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση ισχυρών ρυθμιστικών οργάνων τα οποία θα εποπτεύουν τους εναέριους χώρους, τον εναέριο χώρο στα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι και εδώ πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα και το γνωρίζουμε και από άλλες συζητήσεις, από δίκτυα άλλων επιχειρήσεων. Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός ανεξάρτη... μιας ισχυρής και ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής. Αν υπάρχει αυτή η ισχυρή και ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ε, με διαφορετικό τρόπο πολλά ζητήματα, δημιουργώντας ε, ένα δίκτυο μεταξύ ισχυρών ρυθμιστικών αρχών, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Τι προτείνουμε λοιπόν. Θα τα περάσω πολύ γρήγορα τα 7 σημαντικότερα θέματα. Πρώτον, ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Εθνικής Αρχής Εποπτείας, των Εθνικών Αρχών Εποπτείας και περισσότεροι πόροι να πάνε σε αυτές. Δεύτερον, βελτίωση της ανεξαρτησίας της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στο, στο κομμάτι των επιδόσεων. Τα βλέπουμε αυτά στις συζητήσεις ε, για τους στόχους της δεύτερης περίοδου. Εκεί έχουμε μια πολύ ανάλογη περίπτωση. Τρίτον, να υπάρχει μια εστίαση στους πελάτες εκ μέρους των αρχών εναέριας πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών αρχών διαχείρισης του εναέριου χώρου. Τέταρτον, πρέπει να επιτρέψουμε την καινοτομία, την εξοικονο... τις εξοικονομήσεις κλίμακας, την βελτίωση των επιδόσεων δίνοντας δυνατότητα να δοκιμαστούν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, στις ε, υπηρεσίες υποστήριξης. Και πάλι να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Δεν μιλάμε εδώ για ιδιωτικοποίηση. Ορισμένες από τις υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται από πάρα πολύ αποτελεσματικά ε, κρατικά όργανα και υπηρεσίες. Και ο όρος unbundling ε, που χρησιμοποιείται, αποδέσμευση, είναι λάθος λέξη. Όλοι το ξέρουμε. Unbundling, αποδέσμευση, ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει να ξεχωρίσουμε την παροχή και την, ε, την δημιουργία των υποδομών από την παροχή των υπηρεσιών. Δεν προτείνουμε εμείς κάτι τέτοιο εδώ. Ε, εδώ το όργανο που παρέχει τις υπηρεσίες είναι επίσης το όργανο που είναι αρμόδιο και για την ανάπτυξη των υποδομών. Πέμπτον, ενίσχυση της δυνατότητας ευελιξίας ε, σε αυτά τα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου. Έκτον, ενίσχυση του μάνατζερ των δικτύων έτσι η διαχειριστική αρχή των δικτύων θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και να συντονίζει το εθνικό και το περιφερειακό και το τοπικό δίκτυο και τέλος να επιληθούν τα θέματα διακυβέρνησης τα οποία έχουμε ε, με όλες αυτές τις διαφορετικές αρχές που υπησέρχονται στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, να ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του, του, του Eurocontrol. Το Eurocontrol εστιάζει στα λειτουργικά ζητήματα μέσω ενός ε, διαχειριστή του δικτύου. Ε, ε, ο, φορέας, ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ασφάλειας, EAA, θα έχει την ευθύνη σύνταξης και εποπτείας της υλοποίησης όλων των τεχνικών κανόνων αεροπλοείας και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εστιάζονται στην πολιτική και στις οικονομικές ρυθμίσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα 7 θέματα τα οποία ε, ε, συμπεριλαμβάνονται στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Οργανισμό 2 ΣΥΝ. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια πολιτική που εισαγάγουμε. Ε, Όλοι τι κάνουμε έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής μας και σκοπό έχει να διορθώσει τα κακό κείμενα της προηγούμενης πολιτικής μας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άτυπο συμβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαϊνέσκο, ο οποίος συμμετείχε στο Βίλνιους σε αυτό το άτυπο συμβούλιο, όπου διαπιστώσαμε ισχυρές αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη κατά της πρότασής μας. Ε, ιδιαίτερα, ε, ε μα, ιδιαίτερα όσο αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης. Όταν έφυγα από εκείνο το συμβούλιο, είπα στον εαυτό μου, τέλεια, έχουμε την δέσμευση όλων των Υπουργών να εφαρμόσουν τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2 συν, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Γιατί ε, αυτή ήταν και η αντίρρησή τους. Δεν θέλουμε το κάτι καινούριο, αλλά θα υλοποιήσουμε τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Εμείς θα τους ελέγξουμε. Και σας χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε ε, τη δική σας δράση για να εξασφαλίσετε ότι, το, ότι ο, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός 2 συν θα βελτιωθεί και σας καλώ να μας βοηθήσετε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια και να βελτιώσουμε τα θέματα αυτά τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σαφείς δηλώσεις σας. Τώρα θα ακούσουμε τους συναδέλφους. Ξεκινάμε από τον κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή για αυτήν την ε, παρουσίαση. Είναι σαφές ότι δεν έχει συμβεί τίποτε το θεαματικό την τελευταία πενταετία από τότε που εγκρίθηκε το δέσμη μέτρων για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό στη δεύτερη φάση του. Δεν έχουν κάνει τίποτα ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη για να πετύχουν να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ούτε σε επίπεδο χάβη και αεροδρομίων, κομβικών, τίποτα από αυτά που αναφέρατε. Πολύ γραφειοκρατικό άχθο και πολλά χαρτιά, πολλή χαρτούρα. Κατά την άποψή μου τα μπλοκ ούτε καν χρειάζονται, χάσιμο χρόνο είναι και κοστίζουν και πολύ χρήμα και δεν προσφέρουν τίποτα το νέο, το καινούριο, προκειμένου να δημιουργηθεί όντω ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Το CES, το SES e μάλλον, 2 συν, όπως το είπατε, γνωρίζει πολύ μεγάλη αντίσταση από τα κρατημέλη. Αντιστέκονται Τουλάχιστον έτσι αντιδράει το Συμβούλιο. Δεν θέλουν ούτε καν να διοργανωθεί κάποια συζήτηση και σε κάθε συνάντηση που είχαμε ως τώρα κατανοούμε ότι δεν θέλουν, δεν θέλουν να συζητήσουν ε, ούτε καν την ανάθεση εντολής προς το Κοινοβούλιο. Θέλουν να τα αφήσουν όλο αυτό μέχρι την επόμενη θητεία, μετά τις ευρωεκλογές. Τίποτε μέχρι τον Απρίλιο της ερχόμενης χρονιάς. Είναι περίεργο όμως. Είναι περίεργο που τα επιχειρήματα κατά του SES 2 e ε, έχουν πιο πολύ να κάνουν με τα θέματα δίκησης. Κανείς δεν συζητά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Όλοι συζητούν τα της τη διαχείριση. Τι θα γίνει με τις αρχές, με τους φορείς, με το σχέδιο επιδόσεων. Οι αντιρρήσεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την επίτευξη του ευρωπαϊκού ουρανού. Δεδομένης της τάσης λοιπόν των κρατών όπω όπως είπατε κι εσείς, και λόγω των εθνικών μονοπωλίων, καταλαβαίνω ότι η μόνη δυνατή λύση θα ήταν να έχουμε μια γρήγορη λύση με μια προσέγγιση top-down, από πάνω προς τα κάτω. Θα ήταν καλό να είχαμε κάποια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Και θα ήταν ίσως η μόνη λύση αυτή. Τι καινούργιο φέρνει το SS2 σε σχέση με το προηγούμενο πακέτο. Τίποτε το θεματικό. Κάποια αποσαφήνιση, αλλά δεν υπάρχουν σοβαρά βήματα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός ενίου ευρωπαϊκού ουρανού. Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση αυτή. Και θα ήθελα εντάχει να σας πω τι εγώ πρότεινα και τι σκοπεύω να προτείνω. Υπέβαλα μία έκθεση, αλλά θα υποβάλω και τροπολογίες. Ας ξεκινήσω με την ανεξαρτησία των ε, ε, αρχών ελέγχου, των υποπτικών αρχών. Πιστεύω ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ εθνικών φορέων μεταξύ των εθνικών αρχών, διότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένας φορέας. Διότι ο κανονισμός είναι ένας. Όχι και αρχές παρακολούθησης και αρχές επιτήρησης. Ο κανονισμός διέπει όλες τις εποπτικές ε, ευθύνε για ένα αεροδρόμιο και για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας. Χρειάζεται λοιπόν μόνον μία εθνική αρχή η οποία θα πρέπει να συντονίζεται ή τέλο πάντων να εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή. Εάν δεν γίνουν έτσι τα πράγματα, κατά την άποψή μου, ο Ευρωπαϊκός Φορέας, η Ευρωπαϊκή Αρχή η μόνη ευθύνη που θα έχει είναι να δίνει συγκεκριμένε τεχνικέ προδιαγραφέ. Αλλά όχι να τι υλοποιεί, να ασχολείται με την υλοποίησή του. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε, πιστεύω. Για το διαχωρισμό τώρα, το unbundling, όπως το είπατε. Είναι, ε, νομίζω, πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τέτοιες υπηρεσίες να πούμε ευθύ εξ αρχή ότι η αεροπλοεία και οι τηλεπικοινωνίε πρέπει να διαχωριστούν τελείω από τον έλεγχο ενέργεια κυκλοφορία και τα συστήματά του. Είναι δύσκολο, αλλά έκανα την εξή πρόταση. Οι παρέχοντε τι υπηρεσίε να υποχρεούνται να εξετάζουν προσφορές και από άλλους παρεχόντες υπηρεσίες για την επικοινωνία, για την αεροπλογία, για τις μετεωρολογικές ε, πληροφορίες και το καθεξής, αλλά να μην υποχρεούνται να διαχωρίσουν μεταξύ διαφορετικών εταιριών την ανάθεση, όπως προτείνει και ορίζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των επιδόσεων τα προγράμματα επιδόσεων όπως ονομάστηκαν, οι υπηρεσίες ε, εναέρειας κυκλοφορίας, με συγχωρείτε μάλλον οι παρέχοντες της πληροφορίας, τις υπηρεσίες, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια των επιδόσεων. Θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει εμείς να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνουν να καλύπτουν αυτέ τι απαιτήσει. Αυτή νομίζω θα ήταν μια συμβαστική λύση. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα λοιπόν των επιδόσεων, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει τον τελευταίο λόγο. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι θα πρέπει να τηρούνται και να λαμβάνονται υπόψη όταν ορίζονται οι εθνικοί στόχοι. Η μόνη λύση που έχουμε τώρα ως ενδεχόμενη Δεδομένη της κατάστασης στα κράτη-μέλη, ο μόνος τρόπος που θα μας επέτρεπε να δημιουργήσουμε τον, τον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό είναι να αξιοποιήσουμε τα τεχνολογικά μας μέσα, να εφαρμόσουμε τα συστήματα που έχουμε από τη ΣΕΖΑΡ. Τα συστήματα αυτά έχουν μελετηθεί και έχουν ήδη μπει στην αγορά χάρη στη ΣΕΖΑΡ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να ορίσουμε με σαφήνεια τις ευθύνε, διότι υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί για τη διαχείριση, για τους υπεύθυνους της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών και οι μάνατζερ θα πρέπει να αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνε, να αναλαμβάνουν τις ευθύνε για όλα τα προγράμματα ώστε να υπάρχει απαραίτητο συντονισμός και ο συγχρονισμός όταν μιλάμε για την υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων ταυτόχρονα. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε προβλήματα με, την, ε, τα δεδομένα λόγω χάρη που είχαμε ως τώρα. Η υλοποίηση μπορεί να ήταν κάποιες φορές επιτυχημένη στην εναέρια κυκλοφορία και όχι στο έδαφος. Θα πρέπει όμω να γνωρίζουν οι παρέχοντες τι υπηρεσίε ακριβώ ποιε είναι οι υποχρεώσει του. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι διαχείριση των συστημάτων Σέζαρ και ποιοι ελέγχουν τον εναέριο χώρο. Θα πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι για τον έλεγχο και υπεύθυνοι για την ανάπτυξη. Αυτά είναι τα στοιχεία που ήθελα να παρουσιάσω και να εισαχθώ στην πρότασή μέσα των τροπολογιών μου. Να επαναλάβω αυτό που είπατε κι εσείς, κύριε Γενική Διευθυντά ότι οι στόχοι για την ασφάλεια δεν είναι για την ώρα αρκετοί δεν επαρκούν. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί επαρκώ υπόψη η πτυχή της ασφάλειας. Να επιμείνουμε μάλιστα σε αυτό. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε, βρίσκεται, σε διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη περίοδο των προγραμμάτων επιδόσεων και ελπίζω ότι θα τα καταφέρετε ώστε να μην περιέλθουμε σε κατάσταση ανάλογη με τη σημερινή. Τα unit Trades, βέβαια είναι κάτι που έχει ακουστεί, έχει συζητηθεί, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε το τι θα πρέπει να καταβάλουν οι ε, ε, αεροπορικές εταιρείες το 2014 αναδρομικά για το 2012. Εάν το σκεφτείτε αυτό θα καταλάβετε ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και δεν έχουν γίνει σε καμία περίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και λίγο χρόνο στους κύριους συγκητές. Ο κύριος ε, Σασόνη. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά της και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την ε, διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας και της αεροπορικής υπηρεσίας. Κατά τη δική μου άποψη, εφόσον θέλουμε να υπάρξει εξέλιξη στο ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό της Αεροπορικής Ασφάλειας θα πρέπει να γίνει κάτι. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τέτοια ε, εξέλιξη χρειάζεται και από την πλευρά της ασφάλειας και των προδιαγραφών τη και των απαιτήσεων να γίνουμε πρωταγωνιστές, διεθνείς πρωταγωνιστές σε ένα παγκοσμιωμένο πλέον σκηνικό. Όλο ένα και πιο ενιαίο. Χωρίς όμως να μπούμε στις ε, λεπτομέρειες του κειμένου, κείμενο που υποβλήθηκε στις 14 Νοεμβρίου, λέει ο μιλητής, στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχουμε πάντως μια μεγάλη ε, ευκαιρία να αλλάξουμε το πώς ε, λειτουργεί ο οργανισμός, αξιοποιώντας και τον τη διαθεσμική συμφωνία για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών του Ιουλίου του 2012. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν καταλήξει σε μια κοινή προσέγγιση για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Μιλάμε για μια συμφωνία που δεν είναι μεν δεσμευτική, από νομικής όμως πλευράς βασίζεται σε μια αναπερίπτωση προσέγγιση. Υπάρχουν βήματα προόδου σε πολλές μα πολλές πτυχές. Δημιουργία οργανισμών, επιλογή της έδρας, ε, governance, διαχείριση δηλαδή, ε, λειτουργία, χρήση των πόρων και διαδικασίες ελέγχου. Πρωταρχικός στόχος του κανονισμού που τώρα εξετάζουμε είναι να ορίσει και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο και ομοιόμορφο επίπεδο για την ασφάλεια της αεροπλοείας, της πολιτικής αεροπλοείας στην Ευρώπη και να δημιουργήσει την απαραίτητη δομή και σύστημα διαχείρισης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να περάσει σε ανακατανομή των ε, αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΑΖΑ και Eurocontrol προκειμένου η ΕΑΖΑ, δηλαδή αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, να ασχοληθεί με την ε, σύνταξη και την παρακολούθηση του πώς υλοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές για την αεροπορική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον οικονομικό σκέλος, ενώ ο Eurocontrol με τη λειτουργική πτυχή όπως διοργανώνεται βάσει της αρχής του φορέα διαχείρισης του δικτύου. Κατά την άποψή μου πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΑΖΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί τελικά ένας φορέας ο οποίος εν τέλει θα αναγνωριστεί ως κατεξοχήν συνομιλητής όλων των ενώσεων, όλων των υπήρων Δηλαδή θα υπάρχει μια δομή πραγματικά διεθνής. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η ΆΖΑ έχει συνάψει σοβαρές ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης με χώρες όπως ε, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, το Ισραήλ και αυτό βεβαίως θα ωφελήσει. Θα είναι ένα ατού και για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τις καλές πρακτικές που ελπίζουμε ότι θα φέρουν ωφέλη σε όλους. Σε ό,τι αφορά το κόστος, το κόστος λειτουργίας του οργανισμού, και εδώ θα ολοκληρώσω, είμαι πεπισμένος ότι το κόστος δεν πρέπει να αυξηθεί, διότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα αλυσιδωτός, θα δημιουργηθούν αλυσιδωτές επιπτώσεις για τις υπόλοιπες για τους υπόλοιπους οργανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε τα θετικά αυτά εργαλεία που θα μπορέσουν να επιτρέψουν την καλή λειτουργία του οργανισμού χωρίς αύξηση του κόστους λειτουργίας του. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. κύριος και ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας, από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχετε τρία λεπτά για να μας πείτε την απόψή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα για τον ε, ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2 ΣΥΝ. Έχουμε ετοιμάσει πολλά κείμενα το τελευταίο διάστημα, αλλά στην δική μας την Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι η ευκαιρία της συζήτησης της σημερινής είναι πολύ επίκαιρη. Έχει γίνει αποδεκτό το πακέτο αυτό, μεν, αλλά αν δείτε τη στάση των κρατών μελών, αντιμετωπίζουν σαν να είναι κάτι επικίνδυνο. Δεν μπορεί το σύστημα αυτό να αντιμετωπίζεται σαν κάτι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τις αερομεταφορές, δηλαδή την κινητικότητα. Είναι μέρος της όλης διαδικασίας και αυτό. Το ATM αλλά και η SNSP δεν είναι η κάτοχοι του εναέριου χώρου. Πρέπει το σύστημα να γίνει ανταγωνιστικό. Θα πρέπει να δούμε ότι κάποιες φορές λειτουργούν ε, ξεχωριστά τα δύο αυτά συστήματα και οι φορείς. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, γιατί είναι ένα βασικό σφάλμα. Αν δείτε τώρα τις συνθήκες της ευρωπαϊκής αεροπλοείας, ιδίως τι γίνεται με τον τελικό χρήστη που είναι οι αεροπορικές εταιρείες, είναι χάλια η κατάσταση. Είμαστε από τι λιγότερο ανταγωνιστικέ εταιρείε στον κόσμο όσο αφορά την αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι υπάρχουν και οικονομικοί φορεί οι οποίοι θα πρέπει να είναι βιώσιμοι. Εάν δεν είναι βιώσιμοι, τι κινητικότητα θα έχουμε τελικά στην Ευρώπη. Η Επιτροπή μα λοιπόν ήθελε να τονίσει τα εξή σημεία εντάχει. Πρώτα απ' όλα λέει για το ε, σύστημα του ενίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΣΥΣ 2 συν ότι είναι από τα πληρέστερα συστήματα για τη δημιουργία τη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στον εναέριο χώρο. Δεν πρέπει τα κάτι μέλη να σταθούν εμπόδιο σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι λογικό. Και σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ATM, δεν υπάρχει λόγο να μην ακολουθήσει τι βέλτιστε πρακτικέ τη αγορά. Αλλά πρέπει να είναι και αποτελεσματικό. Γιατί να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ATM ε, που να διαφέρει πάρα πολύ από ό,τι η SNSP και να μην ακολουθεί τα πρότυπα της ε, αγοράς στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του συστήματος, θα συμφωνήσω με τον ε, Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε ταχύτητα και πάρα πολλοί στόχοι τώρα δεν έχουν επιτευχθεί. Πολλά είναι τα κράτη-μέλη που έχουν τιμωρηθεί γιατί δεν ε, επιδίωξαν τους στόχους όπως έπρεπε και αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας περισσότερο top-down, από την κορυφή προς τα κάτω δηλαδή, και να δούμε κατά πόσον είναι δυνατή η αποσύνδεση των υπηρεσιών, το unbundling. Και βεβαίω τι θα γίνει με του χρήστε του ενέργειου χώρου. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά πόσον μπορεί να ε, αναθεωρήσει τη σύμβαση για να παίξουν καλύτερα το ρόλο τη η ε, και ελπίζουμε και το Ευρωκοινοβούλιο εδώ να αναλάβει πλήρω το ρόλο που του αρμόζει και του αναλογεί. Σα ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με του συναδέλφου. Γιατί και ο χρόνος πιέζει, νομίζω το πολύ δύο λεπτά στον κάθε ομιλητή. Γιατί και ο κύριος Ζωρίτ πρέπει να μπορέσει να αντιδράσει. Ο κύριος Δανέλη. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Ε, η σημερινή κατάσταση με 28 διαφορετικά εθνικά συστήματα υπηρεσιών αεροναυτιλίας και πάνω από 60 ε, κέντρων ελέγχου ε, είναι προφανώς ε, επιζήμια διότι επιβαρύνει τους επιβάτες με επιπλέον κόστος και καθυστερήσεις διότι δημιουργεί ζητήματα πολύ έντονα επιχειρησιακά και οικονομικά στις αεροπορικές εταιρείες και ευθύνεται βεβαίως για υπολογίσιμου μεγέθους εκπομπές άνθρακα. Άρα τίθεται το εύλογο ερώτημα γιατί τα κράτη μέλη αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο στην εφαρμογή. νομίζω ότι ο λόγος είναι πολύ απλός γιατί στο συγκεκριμένο τομέα έχουμε να κάνουμε με ένα δημόσιο μονοπόλιο το οποίο συντηρείται με ιδιωτικά κεφάλαια και μέσω αυτής της διαδικασίας νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα αυξημένο προστατευτισμό σε κλειστούς επαγγελματικούς κλάδους με συγκεκριμένα και εκτιμένα συμφέροντα και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ε, συνοδεύεται από τη συντήρηση κάποιων ιδεολειψιών του παρελθόντος σχετικά με εθνικές καχυποψίες. Και αυτά βεβαίως είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό νομίζω ότι η εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού ε, έχει ένα ισχυρό ε, ενωσιακό, συμβολικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, πέρα από τα πρακτικά ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Ε, θέλω να υποβάλω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Θα τις κάνω όσο γίνεται πιο σύντομες. Σχετικά με το νομικό διαχωρισμό των υποστηρικτικών υπηρεσιών, η εμπειρία από άλλους τομείς, όπως είναι στους σιδηροδρόμους κυρίως, μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλές, πολύ μεγάλες δυσκολίες στην υλοποίηση. Ε, η πηγή του προβλήματος δεν είναι ότι είναι ανεξάρτητες δεν είναι ανεξάρτητε οι υπηρεσίε. Νομίζω ότι είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τι υποχρεώσει του. Ε, αν λειτουργήσει καλύτερο μηχανισμός επιδόσεων ή αν τεθούν ειδικοί στόχοι για τις ε, υποστηρικτικές υπηρεσίες, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να επιβληθεί διαχωρισμός στους πάντες. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι όσον αφορά τα μέτρα για τις εθνικές εποπτικές ε, αρχές, που είναι ό,τι σημαντικότερο για την υλοποίηση του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού, νομίζω ότι αν δεχτούμε ότι θα πετηθούν 7 χρόνια, για 7 χρόνια δεν θα γίνει τίποτα ουσιαστικά διαφορετικό από αυτό που σήμερα ισχύει. Άρα νομίζω πρέπει να συντομευθεί ο χρόνος αυτός. Και τέλος, ο κλάδος ο συγκεκριμένο με όλα τα παρακλάδια του και οι εργαζόμενοι θα υποστούν πολύ μεγάλες πιέσεις στα επόμενα χρόνια, όχι τόσο από την υλοποίηση του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού, όσο από τις τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες έρχονται. Ε, έτσι λοιπόν νομίζω ότι αφού χαράσουμε κοινοτικούς κανόνες ε, για την οικονομική και επιχειρησιακή λειτουργία του κλάδου, οφείλουμε να χαράξουμε και κανόνες και μέτρα για την αξιοποίηση και προστασία έτσι ε, έμεσα βεβαίως για το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Ε, συμφωνείτε ότι θα πρέπει να υπάρξουν και τέτοιες βλέψεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ κατάλαβα πως ο κύριος Γκρός θα παρέμβει, έτσι. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Ε, έχω την αίσθηση ότι τα έχω ξαναδεί όλα αυτά, όλη αυτή τη συζήτηση. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, την οποία δεν τηρούν. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αυτό. Η υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχει. Μπορεί να βελτιωθεί με την ε, πρόταση αυτή, αλλά δεν αλλάζει η κατάσταση. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν στη μεταβατική φάση. Υπάρχουν οι χώρες με αρνητική και παθητική στάση. Θα τις αφήσει ίσχυση ή θα ακολουθήσει κάποια άλλη διαδικασία για να ασκήσει κάποια πίεση. Γιατί για εμένα είναι απλό. Είτε αποδεχόμαστε την ε, κατάσταση, την τωρινή, κάτι νέο. Δεν μπορεί να μην έχουμε τίποτα. Η αιτιολόγηση τότε δεν μπορώ να την καταλάβω εγώ ούτε οι πολίτες. Δηλαδή αν θέμε, αν μπορούμε να είμαστε ασφαλέστεροι, αποτελεσματικότεροι, πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και φτηνότεροι, δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουμε το σύστημα. Και δεύτερο ερώτημα, ξέρουμε ε, πόσο σημαντικά εμπόδια υπάρχουν στις χώρες, αναφέρθηκαν, το ανθρώπινο κεφάλαιο που υπάρχει πρέπει να διατηρηθεί, Βεβαίω το ανθρώπινο κεφάλαιο ε, έχει και κάποιο κόστος. Η Κομισιόν θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα. Δεύτερον, για κάποιες χώρες είναι σημαντικότερο το θέμα των εσόδων, ε, σημαντικότερο από το θέμα της συνεργασία. γιατί και τα έσοδα είναι σημαντικά. Ε, είδαμε το απλό παράδειγμα του, του Μάστριχτ, πώς δόθηκαν δηλαδή κάποιες ε, απαντήσεις. Εάν γνωρίζουμε αυτές τις αδυναμίες, νομίζω πως μπορούν να αναφερθούν σε αυτήν εδώ πέρα την πρόταση. Κάτι ακόμα, ε, μπορούσα να πω πολλά, αλλά θα αναφερθώ μόνο σε αυτό. Είναι και χωρισμένος ο αέριος χώρος μεταξύ της ε, ασφάλειας του επίπεδου του κράτους και της ανέρειας κυκλοφορίας. Η Κομισιόν θα το δει αυτό το θέμα προληπτικά, γιατί αν δούμε τι γίνεται στην κεντρική Ευρώπη και το τι απομένει από πλευράς ένα αέριου χώρου, τίθεται και ζήτημα ασφαλείας ε, πλέον. Τέλος, και μια απλή ερώτηση. Νομίζω είχαμε και την έκθεση του συντονιστή του κυρίου Γιάννη που την διαβάσαμε. Βεβαίω ως ε, συντονιστή ήταν κάπως πιο διπλωματικός από ότι ω ε, βουλευτής, αλλά σαφές είναι δεν το θέλουν οι χώρες. Οπότε το ερώτημά μου είναι, ποιο ε, επιχείρημα έχετε για να είστε πιο αισιόδοξο ότι θα πείσετε τις ε, χώρες. Ε, υπάρχει εδώ πέρα κάποιος πίσω από την πόρτα που εμποδίζει, είστε πιο ε, θετικός τώρα. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα και τις κυρίες. Η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ. Κύριε Φαντάλεν. Θα είμαι και πιο σύντομη από τα δύο λεπτά. Ο Ματιέ ανέφερε κάποια πράγματα. Πράγματι, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπαμε όλοι πως δεν είναι δυνατόν να χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό εναέριο χώρο που θα είναι πιο αποτελεσματικός, ε, να το υπογράφουν όλα τα κράτη-μέλη και να μην εφαρμόζουν τίποτα. Γι' αυτό α, αντιλαμβάνομαι την Κομισιόν που έκανε μια πρόταση απόρρισα που τα κράτη-μέλη είπαν πως ε, ε, θα πρέπει να έρθει πιο γρήγορα η πρόταση για να την εφαρμόσουν. Γνωρίζω βεβαίω πω ε, τα κράτη-μέλη έχουν πάρα πολύ διαφορετική οργάνωση όσον αφορά τη διαχείριση του εναερίου χώρου. Και αυτό δημιουργεί και τα προβλήματα. Ξέρω πώ υπάρχουν προβλήματα μεταξύ ε, Γαλλίας και Γερμανία ήδη. Απλά δεν μπορεί να μην ε, έχουμε τίποτα. Το θέμα λοιπόν είναι τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν εάν είναι πιο δυναμική η πρόταση θα κινηθούν τα πράγματα. Αναφέρθηκε επίσης το ζήτημα του ανθρωπίνου κεφαλαίου και εκεί πέρα υπάρχουν εργαζόμενοι στον τομέα αυτών και πρέπει να ξέρουμε πραγματικά αν είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όπως θέλουμε το ζήτημα προκύπτει το εάν κάθε κράτος μέλος θα διατηρήσει την υπηρεσία του ή όχι ή είναι αποτελεσματικότερη η συνεργασία, μια κατανομή της εργασίας και εδώ πέρα είναι οι δυσκολίες και τέλος αναφέρθηκε η αποσύνδεση το ξέρουμε από τους σιδηροδρόμους και εκεί πέρα προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε ποιο κράτος μέλος έχει ποιο σύστημα και ποια μπορούν να, θεωρούν, να θεωρηθούν υποδειγματικά για να μεταφερθούν στον ευρωπαϊκό χώρο και πρέπει να το κάνουμε αυτό νομίζω και εδώ πέρα περισσότερο από ό,τι τώρα και τέλος Έχουμε ήδη συνεργασία. Γνωρίζω π.χ. μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Υπάρχει. Ίσως πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ε, τελικά χρειάστηκα δύο λεπτά. Τέλος πάντων τελείωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τζάκι Φόρστερ τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε. Ευχαριστώ την Επιτροπή που ήρθε. Ε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο, τον κύριο Μαρινέσκο, αλλά και την Επιτροπή. Ε, ο κανονισμός αυτός για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ήρθε και τον υποστηρίξαμε και εμείς και η Επιτροπή μας και ολόκληρο το Κοινοβούλιο και πριν από δέκα χρόνια όταν Επίτροπος ήταν η κυρία Παλάσιο. Όλα έχουν να κάνουν με την πολιτική βούληση. Όλοι κατανοούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν οι μεγάλες υποδομές και δομές. Δεν θα το αποκρύψω. Είμαι ευρωσκεπτικίστρια, αλλά δεν βλέπω να υπτίθεται κάποιο θέμα εθνικής κυριαρχίας ως προς τον αέριο χώρο. Και μπορώ να σας το πω και εκφράζοντας ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι είναι υπέρ του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, γιατί αυτό είναι μέρος ενός πακέτου. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα δίχως το άλλο. Είμαστε κατασκευαστές, κατασκευαστές υψηλής τεχνολογίας. Θέλουμε να απολύσουμε τα προϊόντα μας σε όλο τον κόσμο. Ανταγωνιζόμαστε τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή μα. Πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω υπάρχουν 28 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και ακόμα και αυτά που ήρθαν ε, πριν έχουν συνυπογράψει γι' αυτό. Ε, ήρθαν μετά από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού έχουν συνυπογράψει, δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, διαπλεκόμενα συμφέροντα και θέσεις εργασίας ε, κτλ. Αλλά ασχολούμαστε τώρα με, με μακρόπνοα πράγματα, ε, με πράγματα που χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Το βασικό όμως είναι να δούμε τους πελάτες. Αυτό είναι πραγματικά. Ε, γιατί ε, οι καταναλωτές μας εδώ στην Ευρώπη πληρώνουν υψηλότερες τιμές για τα εισιτήρια. Ε, ανταγωνιζόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο και δεν κάνουμε τίποτα. Αν θέλουμε να έχουμε πιο απευθείας δρομολόγια, αν θέλουμε πιο αποδοκτική χρήση της ενέργειας, πρέπει να είμαστε πιο πραγματιστές και πρέπει να δούμε τι έγινε με την ιδιωτικοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Όπως είπε και ο Επίτροπος, μπορεί να γίνει μέσω του δημόσιου τομέα, μπορεί να γίνει μέσω της ιδιωτικοποίησης, μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν υπάρχει ένας και μόνο τρόπος. Τα κράτη-μέλη όμως πρέπει να το κινήσουν το θέμα. Πρέπει κάτι να κάνουν. Όλοι χάνουν το χρόνο τους διαφορετικά. Ε, αν μου επιτρέπετε, όσο αφορά την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου, ορισμένες χώρες κάνουν αυτή την ευέλικτη χρήση εδώ και δεκαετίας. Ε, στην αρχή ήταν ε, μόνο τα στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά μετά μεταφέρθηκε το θέμα και στο, στην πολιτική αεροπορία. Τα κράτη, πολλά κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν ούτε στην πολιτική αεροπορία ή στη στρατιωτική αεροπορία να, να, βρουν τρόπους να αλαφρύνουν την συμφόρηση. Συγγνώμη, Πίτερ, ε, το είπαν, τα συζήτησαν οι σοσιαλιστές. Το, ξέρω, Τζάκι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρία λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα τελείωνε. Θα τελειώσω σε ένα λεπτό. Ε, υπήρξε η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, η οποία έτυχε της υποστήριξης του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι τα θέματα που τέθηκαν είναι σημαντικά και θέλω από την Επιτροπή να μάθω πώς θα σμπρώξετε το θέμα αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πια άλλος χρόνος, να χρονο... δεν έχουμε την πολυτέλεια να χρονοτριβούμε, γιατί είναι πολύ υψηλό το κόστας για τις επιχειρήσεις. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρούτε, ακούσαμε κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια. Έχουμε 10 λεπτά, μπορείτε να κάνετε τα σχόλιά σας γιατί 12.30 βεβαίω θα διακόψουμε. λοιπόν πάντα κατά νου το ρολόι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την συζήτηση. Να ξεκινήσω με κάποια γενικά σχόλια. των κυρίων Μαρινέσκου, Καϊτζακά και της κυρίας Φώστερ. Εδώ πέρα το θέμα είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε για να μπορέσουν να επιζήσουν. Και έχουμε ένα σύστημα το οποίο σε ένα βαθμό είναι δομημένο ε, έτσι ώστε το κόστος είναι πολύ υψηλό, οι εταιρείε δεν ε, βγάζουν κέρδος και κάποια στιγμή κινδυνεύουμε να χάσουμε το ότι η Ευρώπη είναι κόμβος αεροπορικός. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε σε ένα βαθμό ίσως να είναι 12 και 5 πλέον, όχι παρά 5. Αν δείτε τις αναδιαρθρώσεις αεροπορικών εταιριών κτλ. Οπότε αυτό είναι το ουσιαστικό πολιτικό μήνυμα εδώ πέρα. που πρέπει να στείλουμε και στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Μαρινέσκου σωστά είπε πως ε, μάλλον πρέπει να το δούμε από πάνω προς τα κάτω το θέμα. Μια τέτοια προσέγγιση η οποία σε ένα βαθμό θα ξεκαθαρίσει το ποιος κάνει τι, ποιος έχει την κάθε ευθύνη και αυτό ακριβώς είναι ο Ευρωπαϊκός Ενέργειος Χώρος 2 συν. Αναμένω τις τροπολογίες σας για να δούμε το τι μπορούμε και να κάνουμε. Μιλήσαμε για την άσκηση πίεσης, ίσως θέλετε να πάμε λίγο παραπέρα. Ε, άκουσα επίσης και μια συζήτηση την οποία ευχαρίστως θέλουμε να έχουμε για το ποιες είναι ουσιαστικές υπηρεσίες και εσείς μιλήσετε για ναυτιλία και επικοινωνίες. Αεροναυτιλία δηλαδή. Να το δούμε λοιπόν πώς θα το ρυθμίσουμε. Είμαι ανοιχτός ως προς αυτό και καλωσορίζω αυτό το οποίο λέτε πως όσον αφορά το θέμα της απόδοσης, η Κομισιόν πρέπει να μπορεί να έχει την τελευταία λέξη. Για τεχνολογία δεν πιστεύω πως χρειάζεται να προσθέσω πολλά σε αυτά τα οποία είπατε. Συμφωνώ πλήρως με τις ανησυχίες σας όσον αφορά τους στόχους για την ασφάλεια. Κύριε Σασόνη, σας όλοι. Η ανάλυση σας πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση με την δικιά μου. Πρέπει δηλαδή η ΕΑΣΑ να γίνει το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασφάλεια και θέματα περιβάλλοντος και να την ενισχύσουμε. για το κόστος. Να πω το εξής. Μεταφέρουμε από το Eurocontrol στην ΕΑΖΑ διάφορες αρμοδιότητες. Πληρωνόταν μέσω των τελών διέλευση των χρηστών. Εάν δεν βρεθεί ένας τρόπος να πληρώνει ο χρήστης, πρέπει να βρεθούν αυτά από λεφτά των φορολογουμένων. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε λίγο το πώς θα είναι δομημένοι οι μηχανισμοί, γιατί κάποιες αρμοδιότητες, ε, διαχειριστές δηλαδή της ενέργειας κυκλοφορίας, το θέμα της εποπτείας, μεταφέρονται στο control. Ε, μεταφέρονται από το Control στην ΕΑΖΑ, με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω πάρα πολύ αυτά που είπε ο κύριος Κράτσουκ γιατί τα ίδια είπαμε και σωστά τα είπατε και για το τι συνέβη στο Βίλνες. Ο κύριος Δανίλης, το, το, το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει κέρια σημασία και συμφωνούμε όλοι πως πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. μεγάλο μέρος είναι οι ελεγκτές συναέρης κυκλοφορίας. Ε, σαφώς, η γνώση τους. Εάν δείτε το αμερικανικό σύστημα και το συγκρίνετε με το ευρωπαϊκό, δεν υπάρχουν πολύ περισσότεροι ε, ελεγκτές συναέρης κυκλοφορίας στην Ευρώπη από στην Αμερική. αλλά το αμερικανικό είναι πιο αποτελεσματικό και φτηνότερο γιατί ε, είναι διαφορετικά οργανωμένο. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα μείωση του αριθμού των ελεγκτών. Ε, πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει το ευρωπαϊκό σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό. Κύριε Γκρός, διαδικασία επί παραβάση. Έχουμε τη διαδικασία αυτή και θα την ε, χρησιμοποιήσουμε προσεχώς παράλληλα με τη συζήτηση για τη νέα νομοθεσία. Αλλά νομίζω πως είναι το μοναδικό άλλο όπλο που έχουμε σε αυτό το πλαίσιο όσον αφορά τα μπλοκ, τα λειτουργικά μπλοκ, το καστό απόδοσης να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την διαδικασία παραβάση. Ξέρετε πως ο Κάλλας, ο, ο Επίτροπος, ο κύριος Κάλλας εδώ πέρα ε, είναι πάρα πολύ δραστήριος ε, όσον αφορά τώρα την διανομή κατανομή του αέριου χώρου Μιλάμε για μια, δεν ξέρω πώς είναι στα γερμανικά, μια ενισχυμένη ευελιξία στη χρήση του εναερίου χώρου. Δηλαδή ακόμη περισσότερο από, το, από ό,τι τώρα. Είναι ήδη ευέλεκτος ο αέριο χώρος. Πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο αυτό. Και βέβαια εδώ πέρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το Eurocontrol και η ενίσχυση της λειτουργίας του Eurocontrol ως ε, ε, διαχειριστή του δικτύου. Η κυρία Να ξεκινήσω από το τέλος. Συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Με τον ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2 κάναμε το λάθος πως ε, αυτό είναι το σύστημα και τώρα πρέπει να συνεργαστείτε είτε θέλετε είτε όχι. Αυτό το οποίο προτάνουμε στον Ιερό Ευρωπαϊκό Ουρανό 2 συν είναι ακριβώς η ευελιξία. Δηλαδή πάνω και δίπλα από την δομή των, α, των ΦΑΠ να έχουμε κάτι άλλο εάν έχει νόημα. Ναι, αυτό ακριβώς κάνουμε. Στα υπόλοιπα ερωτήματα νομίζω απάντησα. Για την κυρία Φώστερ. Καταλαβαίνω τι είπατε, πράγματι. Και καμιά φορά απογοητεύομαι κι εγώ, όσο κι εσείς, για το ότι δεν κάνουμε τίποτα. Να πω το εξή. Αυτό που προσπαθούσα να πω είναι πως πραγματικά παλεύουμε και δεν είναι ικανοποιητικά τα πράγματα, αλλά υπάρχει κάποια κινητικότητα και είδαμε κάποια βελτίωση. Εσείς λέτε πως το ποτήρι είναι άδειο. Εγώ θα έλεγα πως πάντα είναι μισογεμάτο. Εγώ το βλέπω, πρέπει να το γεμίσουμε τώρα μέχρι πάνω. είναι δυτή η προσέγγιση δηλαδή κάνουμε και προτάσεις και ταυτόχρονα κινούμε διαδικασίες ε, επί παραβάση. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας εκθέσατε τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την υπομονή σας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Τρεις και μισή. Συνεχίζουμε με τη μήνυ ακρόαση. Καλή σας όρεξη.